Συνάδελφοι, να καθίσετε, παρακαλώ, και όποιοι δεν ε, είναι προσκεκλημένοι ή δεν ε, μπορούν να παρίστανται σήμερα, ε, παρακαλώ να αποχωρήσουν, να βγουν εκτός αθούσης. Ε, να καλωσορίσω τον ε, Επίτροπο Έτινγκερ, είναι μαζί μα σήμερα για να δούμε τα θέματα τη ενεργειακή πολιτική. Θα ακούσουμε λοιπόν πολλά ενδιαφέροντα από τον ίδιο και θα δούμε τι γίνεται με την ενεργειακή πολιτική, ποια είναι τα μεγάλα project που έχουμε μπροστά μα. Οπότε παρακαλώ να τον ακούσετε προσεκτικά για να θέσετε μετά ερωτήσει. Έχουμε μέχρι τι 4 καιρό γιατί μετά θα έρθει ο επόμενο επίτροπο. Herr Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας για το 2012. Η Επιτροπή θα σας αναφέρει τι ακριβώ γίνεται με την ενεργειακή πολιτική, η οποία θα αποτελέσει πάλι σημαντικό κομμάτι τη ε, πολιτική μα. Η ενέργεια στο πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής αποτελεί ψηλή προτεραιότητα. Θεωρούμε ότι δεδομένε και της κρίσης και για να επιτύχουμε την ανταγωνιστικότητα τη οικονομία μα, αλλά και προ όφελο των καταναλωτών μα, πρέπει να έχουμε κοινή, ευφυή ενεργειακή πολιτική και να εξευρωπαίσουμε την ενεργειακή πολιτική κάτι που θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική βάση, εάν επιτευχθεί. Μια, ένα, μια σύντομη αναδρομή του περασμένου έτους. Τι κάναμε μέχρι τώρα, τι καταφέραμε, τι έγινε με τις διαβουλεύσεις μας. Καταρχάς, βρισκόμαστε στην αποφασιστική σημασία φάση για την ε, ενεργειακή απόδοση. Η πρόταση υπάρχει για μια νομοθεσία με μια ε, δύο βαθμίδων στρατηγική. Υπάρχουν δεσμευτικά μέτρα που έχουν υποβληθεί και ευχαριστώ για την ε, συνεχή ε, υποστήριξη που μας δίνει το Κοινοβούλιο, ε, κάτι που προκύπτει από όλα τα κόμματα, από όλες τις πολιτικές ομάδες. Εσείς λοιπόν είσαστε αυτοί που μας κινείτε και όσο πιο πολύ μας υποστηρίζετε, τόσο πιο α, πολύ μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Η θέση των α, κρατών μελών βεβαίως στο Συμβούλιο είναι πάντα αρκετά διαφοροποιημένη, πολύ ετερογενής και ελπίζουμε η νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση κατά τη διάρκεια της ε, Δανεικής Προεδρίας να μπορέσει να, έχει, ε, να αποφέρει αποτελέσματα μέχρι τον Ιούνιο. Επίσης, προχωράμε πολύ καλά στο θέμα των ε, δικτύων και των υποδομών. Έχουμε την νομοθεσία για μια επιταχυμένη διαδικασία αδειοδότησης και για τη συγχρηματοδότηση υποδομών καθώς επίσης έχουμε και την πολυετή πρόταση της Κομισιόν για τον, για τον προϋπολογισμό Έχουμε το Connecting Europe Facility που έχει συγκεκριμένη πρικοδότηση από τον προπολογισμό και επίσης έχουμε την εξωτερική ενεργειακή πολιτική και εκεί έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και βρισκόμαστε σε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με το Κοινοβούλιο για το πώς η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής θα μπορέσει να γίνει καλύτερη στο μέλλον. Επίσης, η ασφάλεια των ε, offshore. Και εκεί υπάρχει πρόταση, εδώ και κάποιες εβδομάδες, συγκεκριμένη. Τελευταίο σημείο για, σε ό,τι αφορά την αναδρομή αυτή. Αλλά και για τις προοπτικές που έχουμε. Τα stress tests που έχουμε κάνει για, τις, ε, για τα πυρηνικά εργοστάσια που υπάρχουν στην Ευρώπη. Η πρώτη βαθμίδα ήταν η, τα τεστ αυτά των ε, ενεργειακών επιχειρήσεων. Τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση με την ε, παρέμβαση και των ε, Υπουργείων και των αρμοδίων ε, υπηρεσιών. Επίσης θα υπάρξει και μια ενδιάμεση έκθεση, η οποία θα υποβληθεί τον Ιανουάριο. Και από τον Ιανουάριο και μετά θα ξεκινήσουν οι αξιολογήσεις ομοτήμων, τα peer reviews και τα ευρωπαϊκά stress tests. Και υποθέτω ότι τα stress tests αυτά δεν θα αποτελέσουν ε, ε, αυτοματισμό σε ό,τι αφορά τις, ε, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ούτε θα μπαίνει αυτόματα από ένα stress test η σφραγίδα ασφαλείας σε μια, σε μια πυρηνική εγκατάσταση. Ας πούμε, η πυρηνική ασφάλεια για την Γαλλία. Πριν από λίγες μέρες υπήρξε μια ενδιάμεση έκθεση η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και λέει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Έχουν γίνει εκεί προτάσεις για το πού και το πώς μπορούν να γίνουν τεχνικές αλλαγές απαραίτητα μετά από τα stress tests. Δείχνουν λοιπόν τα τεστ αυτά ότι ο στόχος είναι ε, μια μεγαλύτερη ασφάλεια για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Τώρα, για την επόμενη χρονιά, το 2012, και το πρόγραμμα εργασίας μας. Το Δεκέμβριο, όπως έχουμε ανακοινώσει, θα υποβάλουμε την πρότασή μας για έναν ε, εργειακό χάρτη για το 2015. Αυτός ο χάρτης θα αποτελέσει μια πρόσκληση. Θα περιλαμβάνει διάφορα σενάρια. θα, έχει, θα αποτελεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική με συγκεκριμένα ε, σημεία για το πώς μπορεί να, έχει, να είναι η πολιτική μας για την ενέργεια μέχρι το 2030. Δεν ε, προκαταλαμβάνουμε τα πράγματα. Ξεκινούμε μια διαδικασία η οποία βεβαίως θα συνεχιστεί. Το 2002 ξεκίνησε η διαδικασία αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια κοινή ενεργειακή πολιτική και πολιτική για το κλίμα. Πέντε χρόνια αργότερα ξεκίνησε ο στόχος 20-20-20 για το 2020. Μία παρόμοια διαδικασία θέλουμε τώρα επί τη βάση αυτών των διαφόρων σενάριων να την ξεκινήσουμε στο Κοινοβούλιο, στα κράτη-μέλη, στην ενεργειακή κοινότητα, στους διάφορους επενδυτές, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όλοι θα συμπεριλαμβάνονται και θα συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. και ελπίζουμε το 2014 και όχι το 2017 να, έχουμε σε, να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα δεσμευτικά αποτελέσματα, ε, προβλέψει για, την επόμενη δεκαετία, α πούμε μέχρι το 2030, και θα έχει βεβαίω και μια μακροπρόθεσμη προοπτική μέχρι το 2050. Έτσι ώστε να έχουμε μέχρι τότε μηδενικέ ε, εκπομπέ ε, διοξιδίου του άνθρακα. Και βεβαίως θα υπάρξουν πολλά σενάρια τα οποία θα συζητηθούν εκτενώς. Ναι. Πέραν του οδικού αυτού χάρτη, θέλουμε να τονίσουμε και την εσωτερική αγορά της ενέργειας. Θέλουμε να σας δείξουμε πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της ε, ενιαίας αυτής αγοράς πού βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει προβλήματα, τι γίνεται με το δεύτερο και το τρίτο πακέτο για την ιστορική αγορά. Θέλουμε να σας δείξουμε επίσης ε, από την επόμενη χρονιά πώς θα εξελιχθούν οι νέες ε, πηγές ενέργειας και πού υπάρχει ανάγκη να συντονιστούμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πρόθεσή τους. Υπάρχει και ένα το ε, πρόγραμμα Ήλιος για την Ελλάδα και πώς δηλαδή μπορεί η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας και τα συστήματα ε, επιχορήγησης των ε, κρατών μελών να συνδεθούν με το πρόγραμμα αυτό. Θέλουμε να τις πηγές ενέργειας, μιλούμε και για τη Βόρεια Αφρική και πώς όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν με το δικό μας σύστημα. Θέλουμε επίσης να σας υποβάλουμε μία μια πρόταση για το CCS, για την δέσμευση και την αποθήκευση του άνθρακα. Και θέλουμε επίσης να υποβάλουμε, να κάνουμε μάλλον μία αξιολόγηση. Και με συναδέλφους προσπαθούμε να εκπονήσουμε μια έκθεση με συνέπειες από όλα αυτά τα προγράμματα, τις οποίες θα συζητήσουμε βεβαίως μαζί σας. Θέλουμε λοιπόν να σας δείξουμε ότι υπάρχουν, ε, υπάρχει μια πληθώρα σχεδίων, ε, νομοθετικών ε, προτάσεων και μέτρων, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν και να αποφασιστούν τον επόμενο χρόνο και επίσης υπάρχουν και κάποια νέα προγράμματα, κάποιες νέες προτάσεις, οι οποίες θα σας υποβληθούν και ε, υποθέτω ότι η ατζέντα σας και για, το, για την ενεργειακή πολιτική θα είναι πραγματικά γεμάτη. Ελπίζω λοιπόν να είναι επικοδομητικές και την επόμενη χρονιά οι συζητήσεις μας όπως ήταν και το 2011. Σας ευχαριστώ πολύ και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για τις, ε, εάν έχετε ερωτήσεις σας να σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και για τις ε, πληροφορίες σας. Να δούμε λίγο τον κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Δελκαστήγιο έχει το λόγο. Ε, για να δούμε αν δουλεύει. Α, δουλεύει. Ωραία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Μισό λεπτό λοιπόν, διακόπτη. Ε, δύο λεπτά αν θέλετε. Δύο λεπτά αν έχετε. Δύο λεπτά μόνο. Ε, gracias, eh, comisario, por estar hoy aquí explicándonos cuál va a ser eh, los objetivos para... Ευχαριστούμε που μας εξήγησε αυτούς τους στόχους για το 2012, για αυτό το γενικότερο το οποίο σε σχέση με την επόμενη χρονιά. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τώρα που κλείνει αυτή η χρονιά θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι αναπτύξατε τρομερή δραστηριότητα εσεί από πλευρά Κομισιόν που <clears throat> εσείς έχετε το χαρτοφυλάκιό σας ε, στη δική σας, στο δικό σας πεδίο ε, δράσης ε, νομοθεσία όσον αφορά τα ενεργειακά ούτω ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη δέσμη μέτρων υποδομής που είναι πραγματικά τόσο σημαντικό Τώρα για την επόμενη χρονιά μας ε, παρουσιάσατε ένα τοπίο με λιγότερη νομοθετική δράση αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό. Αυτό που θέλω να σας πω είναι τα εξής τρία. Πρώτον, δεν ξέρω αν είναι δυνατόν από τώρα να μας εξηγήσετε το τι γίνεται όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια από ό,τι φαίνεται προβλέπεται να, να, να εξελιχθεί για τα τέλη της επόμενης χρονιάς. Αν μπορείτε να μας πείτε από τώρα τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει Πέστε μας τι προβλέπετε τώρα όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Τι γίνεται με την ε, μεταφορά του, της τρίτης δέσμης ενεργειακών ε, μέτρων. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, διότι αν δεν γίνει αυτό, τότε δεν μπορούν να ακολουθήσουν και τα επόμενα βήματα. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μια ειστέρηση σημαντική σε κάποιες χώρες ε, και επίσης θα ήθελα κατά τρίτον να σας πω τι γίνεται με τις ανανεώσιμες ενέργειες δύο την πρώτα πρώτα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες μελέτες επιπτώσεων από πολλές πλευρές και με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι αποφάσεις, οι προτάσεις, οι προσανατολισμοί που αφορούν την καλύτερη ανάπτυξη και χρήση τέτοιων ε, ανανεωσίμων ε, πηγών ενέργειας να γίνουν με όλη την προσοχή, με όλη την προφύλαξη που επιβάλλεται. Τώρα κατά δεύτερον για το ίδιο θέμα να δούμε αν θα πρέπει να το δούμε και από πλευρά νομοθετική για νέου στόχου που αφορούν αυτέ τι νέε πηγέ ενέργεια και να λάβουμε υπόψη ότι τα κράτη-μέλη σύμφωνα με το άρθρο 194 έχουν την ε, σχετική αρμοδιότητα σε σχέση και με το ενεργειακό παγέτο. Και ακριβώς ε, πρόκειται για διαφοροποίηση που ισχύει τώρα από χώρα σε χώρα. Έχουμε το τόσες διαφορές όσον αφορά το τι θα γίνει ανανεώσιμα, πυρηνικά. Άλλα ισχύουν σε κάθε χώρα μέλος. Οπότε γι' αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θεωρώ ότι για το ενεργειακό μείγμα η αρμοδιότητα θα πρέπει να συνεχίσει να είναι εθνική. Εάν θέλουμε το σύστημα να αποδίδει. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαδουρέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, που ήρθατε να μας δείτε σε σχέση με όλη την ενημέρωση που κάνετε, μας εξηγήσατε όλα σας τα σχέδια για όλα αυτά τα θέματα του χαρτοφυλλοκίου σας. Επίσης, Πρόεδρε, θα πρέπει να τον γνωρίσουμε, όπως είπε και η κυρία Καστίγιο, ότι τα τελευταία χρόνια προχωρήσαμε σημαντικά όσον αφορά την κοινωνική νομοθεσία για τα ενεργειακά. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική μας ομάδα θεωρεί ότι ακόμα, ακόμα τα πράγματα επιτέχονται βελτίωση. Και σε σχέση με αυτό έχω τις εξής ερωτησούλες για να μου πείτε τι πρεσβεύεται. Όπως γνωρίζετε η πολιτική μας ομάδα ανέκαθεν πρέσβευε το ότι είναι σημαντικό να καθορίζονται δεσμευτικοί στόχοι, τόσο ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ενεργειακή επανάσταση αυτή την οποία οραματιζόμαστε ως Ευρωπαίοι. Επίσης θεωρούμε ότι η επίτευξη του στόχου της μείωση των εκπομπών του διοξιδίου κατά για το 2020 είναι ένα πρώτο βήμα για την μεγαλύτερη μείωση εν ώψη του 2050. Αυτό περνάει μέσα από κάποια μέτρα. Μέτρα από ενεργειακής, ε, ε, ε ενεργειακής αποτελεσματικότητας όσον αφορά τα κτίρια. Γι' αυτό Κύριε Επιτροπέ, παρακαλούμε, θα πρέπει να παρουσιάσετε μια αναθεωρημένη πρόταση από αυτού και εκεί να υπάρχουν οι δεσμευτικοί στόχοι που να αφορούν την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των ε, οικοδομημάτων, των κτηρίων. Οπότε γι' αυτό και θεωρούμε ότι η στρατηγική για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια θα πρέπει να περιέχει κάποιου δεσμευτικού στόχου για το 2030. Και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο, ούτω ώστε να προχωρήσουμε προ ε, τέτοιε πηγέ ενέργεια. Επίση, Κάτι άλλο θα σας πω, κάτι το οποίο το έχουμε πολύ συζητήσει στην Επιτροπή μας. Όμως, πρόσφατα έχει μπει στο χρονοτούλαβο, δηλαδή μιλώ για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι η έγκριση εκείνης της, ε, της, της ομάδας Focus όσον αφορά αυτό το ηλεκτρικό όχημα θα βοηθούσε με, με, με, σε σχέση και με Sense Οπότε τελικά αυτό το οποίο κατέληξε είναι μια πρόταση για την τυποποίηση όσον αφορά πάλι αυτά τα ηλεκτρικά οχήματα. Μπα και μπορείτε να μα πείτε τι προγραμματίζει, τι σχεδιάζει η Κομισιόν για αυτό. Τέλος κύριε Επίτροπε, αυτό όλο που σας είπα είναι αυτό το οποίο θέλει η ομάδα μα όμω, Για πετε μας Εσεί Εσείς τι οραματίζεστε. Ποιο είναι για σας το ιδανικό, το ιδιώδε σενάριο όσον αφορά τα ενεργειακά στο μέλλον για εκείνο το ερευνητικό πρόγραμμα για το 2020. Εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντλήσουμε όσο γίνεται περισσότερα από τη δουλειά των ερευνητών μας και έτσι να καταλήξουμε σε ανταγωνιστικότητα και χωρίς να έχουμε και τις εκπομπές της βλαπτικές. Και βέβαια πάντοτε μπορείτε να υπολογίζετε τη βοήθεια τη πολιτική μα ομάδα. Σαν να μας λέτε ότι ο παράδεισος βρίσκεται επί της γης, συνάδελφε. Η κυρία Χόλ έχει το λόγο. Thank you. Thank you, Commissioner. Ευχαριστώ πολύ τον, ε, τον Επίτροπο που ήρθε να μας μιλήσει σήμερα. Θα ήθελα να σας κάνω τέσσερις συγκεκριμένε ερωτήσεις Κυρίε, Κυρία, καταρχά για την οδηγία και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Είπατε πώ ε, ε, τα κράτη-μέλη ε, μπορεί να μην συμφωνούσαν και εσεί υποβάλλατε συγκεκριμένε προτάσει. Στο Συμβούλιο όμω ε, τώρα ε, γίνεται κάποια συζήτηση που βλέπουν τα κράτη-μέλη τι έχει προτείνει η Κομισιόν και ενδεχόμενα να χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία και ίσως ε, τελικά ίσως θα ήθελα να, να έχουν κάτι το διαφορετικό. Η Κομισιόν ε, τελικά θα ήταν ευχαριστημένοι με αυτό το οποίο ζητάνε τα κράτη-μέλη. Επίσης μιλήσατε για τους οδικούς ε, χάρτες ε, για την ενέργεια και για το 2030. Αυτό εδώ θα συμπεριληφθούν και οι στόχοι για τις ανανεώσιμες ανέργειες για το 2030. Και το ρωτάω αυτό γιατί η βιομηχανία, αν θέλετε, θέλει να ξέρει ε, τι θα συμβεί μετά, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα στίχος το 2020 και ο, τομέας, ο διευρυνόμενος τομέας της ανανεώσιμης ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ε, ε, βιομηχανία τώρα που περνάμε την κρίση αυτή στην Ευρώπη και θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί μετά. Επίσης για το συντονισμό των συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας να μας πείτε κάτι παραπάνω. Επίσης, ε, μιλήσατε για κάποιες εκτιμήσεις. Ε, εμείς ακόμα δεν έχουμε πάρει τίποτα. Ε, έπρεπε να είχαμε τις εκτιμήσεις αυτές πριν από μήνες. Και θα ήθελα να μου πείτε εάν και κατά πόσον θα υποβληθούν συγκεκριμένα στοιχεία. Και, εν κατακλείδη, όσον αφορά τα πυρηνικά stress test, θα εξετάζετε με ολιστικό τρόπο τις δοκιμές ασφάλειες και θα λάβετε υπόψη σας συνέπειες όπως οι κλιματικές αλλαγές ή το γεγον... ή συν... Ε, δηλαδή οι κλιματικές αλλαγές που οδηγούν σε ακραία καιρικά φαινόμενα, σε πλημμύρες κτλ. Θα το εξετάσετε και αυτό το παράγοντα όταν μιλάτε για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η κυρία Φόρτ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Εν συντομία, για την οδηγία που αφορά τις ε, πλατφόρμες ε, εξόριξης πετρελαίου offshore. Ε, ξέρω ότι θέλετε όλες αυτές οι πλατφόρμες να λειτουργούν με τον πιο ασφαλή δυνατό τρόπο στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα και αυτή ήταν και η πρόθεση της Επιτροπής όταν συντάσαμε και την έκθεσή μας. Στην οδηγία σας όμως ε, η προτινόμενη νομοθεσία δεν είναι τόσο ισχυρή, αν θέλετε, στον τομέα της ασφάλειας, όπως ε, οι διατάξεις που ισχύουν σε κάποια κράτη-μέλη. Και το γεγονός ε, το ότι έχουμε μια οδηγία και όχι κάποιο κανονισμό, τότε νομίζω ότι δημιουργούμε μια νομική ασάφεια και για τους νομοθέτες ε, και για αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ε, και για αυτούς που εφαρμόζουν τις αποφάσεις. ξέρω κύριε Επίτροπε ότι αυτό δεν είναι η πρόθεσή σας ε, και διαρωτώ με μήπως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να έχουμε μέγιστη εναρμόνιση εκεί που είναι απαραίτητο και μήπως κάποια καθεστώτα είναι πιο ισχυρά αν θέλετε σε κάποια άλλα κράτη-μέλη και αυτά να μείνουν εκεί, οι πιο αυστηροί κανόνες να μείνουν Δηλαδή να μιλήσουμε για εναρμόνιση εκεί που χρειάζεται. Και προφανώς η πρόθεσή σας δεν είναι να αποδυναμώσετε ήδη ισχύουσα νομοθεσία, η κυρία Μπομπίνσκα. Μία σύντομη παρατήρηση. Μέχρι στιγμής γυναίκες μίλησαν μόνο εξ των πολιτικών, διαφορών πολιτικών ομάδων και αυτό δείχνει ότι οι γυναίκες ε, ε, ασχολούνται με την νομοθεσία ενώ οι άντρες διαχειρίζονται μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Λοιπόν, είπαμε ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένο, συγκεκριμένες διατάξεις για να υπάρχει και ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο να λειτουργούν εγώ θεωρώ ότι ούτως ή άλλως στο οικονομικό μας περιβάλλον επικρατεί τόσο μεγάλη ασάφεια ε, και κινδυνεύουμε ε, να μπούμε σε μία περίοδο ταραχών, αναταραχών τέλος πάντων και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς ε, στις προτάσεις μας. Η ερώτησή μου ποια είναι πέρυσι και φέτος στο πρόγραμμα εργασίας σας τονίσατε την σημασία της εφαρμογής. Αυτός ήταν ο βασικός εφαρμογής όλων των κανονισμών. Αυτός ήταν ο βασικός στόχος της Κομισιόν. Της Κομισιόν. Και είπατε ότι κυρίως το τρίτο πακέτο είναι το πιο σημαντικό. Τώρα περνάει αυτό και έχετε υποσχεθεί ότι θα ασχοληθείτε με την εφαρμογή των, ε, διατάξεων, των νομοθετικών ε, εργαλείων, αν θέλετε, που αφορούν την ε, εσωτερική αγορά και την ενέργεια. Θα ήθελα, όπως και για την εφαρμογή του τρίτου πακέτου, να, να μου κάποιους φόβους μου. Διάβασα στον ε, τύπο ότι η κυρία Μέρκελ όταν ε, στα εγγένεια της North Stream σας ζήτησε να δείξετε κάποια ευελιξία απέναντι σε χώρες που δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένες ε, με τις λύσεις που προτείνονται στο τρίτο πακέτο. Σε κάποια ρωσικά μέσα ενημέρωσης διαβάσαμε ότι η κυρία Μέρκελ ζήτησε αλλαγές στο τρίτο πακέτο. Επομένως, αυτό που ρωτάω είναι η θέση σας, ποια είναι η δική σας, πώς το βλέπετε. Dobrý den, pane komisaři. Ε, já se pokusím trochu narušit ten... Χαίρετε. Καλησπέρα κύριε Επίτροπε. Για πέστε μας. Να, που μετά από τόσε τόσε κυρίε και ένα άντρα λαμβάνει το λόγο να σα υποβάλει μια ερώτηση. Βέβαια, ναι, είναι αλήθεια ότι εμεί είμαστε το αδύνατο φίλο. Γι' αυτό και πεθαίνουμε και ποιον από τι γυναίκε. Όμω, όμω, σε αυτήν την επιτροπή τουλάχιστον είμαστε περισσότεροι ή ισχυρότεροι. Τέλο πάντων, παρόλα αυτά, εγώ δεν τρέφω τίποτα άλλο παρά θαυμασμό για τι συναδέλφου τη κυρία. Τέλο πάντων, έχω μια σημαντική ερώτηση προ εσά, κύριε Πίτρο. θα παρατηρήσατε αυτές τις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη και ενώ την ε, ενεργειακή δομή κατάσταση των πραγμάτων. έχουμε βέβαια επαναστατικές αλλαγές τον τελευταίο αιώνα. Το δίκτυο της μεταφοράς ενεργείας γίνεται όλο ένα και καλύτερο. Και αυτό αφορά τις διαφορετικές ενεργειακές πηγές, ενεργειακούς πόρους. Τώρα, καταλάβαμε φυσικά ότι η τεχνολογία είναι όλα ένα πιο σημαντικός παράγοντα για την ενέργεια. Εσείς πώς το βλέπετε, τι τεχνολογικές μεθόδους θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε, κάπως να συντονίσουμε τα δίκτυα μεταφοράς ενεργείας. Nejúspěšnější bys eh, v té μιλάω για το χρονισμό, το timing αυτών των δικτύων. Το καθένα έχει το δικό του timing. Υπάρχει κάτι σαν ανταγωνισμός. Αλλά γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε. Για του χρόνου και για το μέλλον γενικότερα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Τι είδου συντονισμό θα μπορούσε να σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται να αναθεωρηθεί προς αυτή την κατεύθυνση το energy mix το λεγόμενο. Ξέρω ότι ο Φρόιντ είπε ότι κάθε <laughs> ανθρώπινο όν έχει και το και και θηλυκό τμήμα ε, κομμάτι. Αυτή τη στιγμή εκφράζει το θηλυκό μου κομμάτι στη συναπογευματινή μας συνεδρίαση. Κύριε Επίτροπε, μας μιλήσατε για τον οδικό χάρτη για το 2030 και το 2050 θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για το 2020. Τι θα γίνει για τον απολογισμό άνθρακα, και τον άνθρακα ε, στην κοινότητα τα, τα επόμενα 8 χρόνια. Φαίνεται ότι υπάρχει καθυστέρηση και τα πράγματα δεν θα φτιάξουν. Εάν ε, βλέπω, αν και τις... Ε, τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ε, από θερμική ενέργεια και ε, από, τον φυσικό, από το φυσικό αέριο, ε, τα πράγματα με ανησυχούν. Επίσης, δεύτερη ερώτηση αφορά το φυσικό αέριο από τη Ρωσία και την εξάρτησή μας από την Ρωσία και το φυσικό αέριο. Τι θα γίνει και τρίτη ερώτηση για την πυρηνική ενέργεια. Μας μιλήσατε για stress test, για δοκιμασίες αντοχής. Μας είπατε ότι θα έχουν σαν, δεν θα έχουν σαν αποτέλεσμα ούτε την, το κλείσιμο των εγκαταστάσεων, ούτε ένα ε, σήμα ποιότητας. Άρα, ποιε θα είναι οι συνέπειες αυτών, αυτής της δοκιμασίας. Σε τι θα χρησιμεύσουν. Συμμάρχε, κύριε Επίτροπε, ομολογώ ότι σας είμαι θα για το ότι κάνετε ό,τι μπορείτε για την κοινή ενεργειακή πολιτική. Και ότι είστε πάρα πολύ αμερόληπτος για τα διάφορα deal που κλείνουν τα κράτη-μέλη ακόμα και το πιο μεγάλο. όμως ήρθε η ώρα της αλήθεια κάποια στιγμή και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό σας το λέω. Γιατί, διότι τώρα ήρθαμε αντιμέτωποι με αυτή την εκστρατεία της Γκασπρόμ, των μονοπωλίων, των Ρώσων τελικά. Και αυτό πλήσει τα θεμέλια, τις αρχές, τα βασικά στοιχεία του Τρίτου Νοικού Οπότε πάνω σε αυτό θα σας ρωτήσω. Μπα και μπορείτε να προβείτε τώρα σε κάποια δήλωση δυναμική, ξεκάθαρη, ότι θα πολεμήσετε για το τρίτο πακέτο κατά των ε, Ρώσων, κατά κάποιων Γάλλων πολιτικών, κάποιων Γερμανών πολιτικών και δεύτερον. Τι λέτε. Αποκλείεται το South Stream να αποκλειστεί ε, για τους τρίτους και έτσι να μην μπορεί να εφαρμοστεί και πέρα το τρίτο παγκέτο. Σας ευχαριστώ για επόμενη κυρία. Επίτροπε, με μεγάλη μας χαρά σας ε, φιλοξενούμε σήμερα εδώ. Δύο, επίσης αναφέρατε δύο σημαντικά στα οποία θέλω να σταθώ. Πρώτα, πρώτα, ότι προχωρεί, επεξεργαζόμαστε αυτό το τρίτο πακέτο. Έχουμε ένα καινούριο χάρτη πορείας για την ενέργεια και θα καλύψουμε έτσι και το φυσικό αέριο. Και το σχιστολιθικό αέριο, οπότε γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα το χειριστούμε σε σχέση με το ρώσικο αέριο και τι θα κάνουμε με την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Τι θα γίνει με την έλλειψη, με την ενεργειακή παινία του Τώρα θα πρέπει να υποστήριξουμε τους στόχους στην κοινωνία. Κάποιοι θέλουν να χρηματοδοτήσουν να επιδοτήσουν το ΣΥΠΗΝ την κατανάλωση σε άλλε ε, χωρισμένε. Δηλαδή, από πλευρά επιμελητία, τι θα μπορούσατε να κάνετε για αυτή την προσπάθεια, την νέα τάση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάτι για την οδηγία τη αποτελεσματική χρήση τη ενέργεια. Από όσο γνωρίζω, δεν θέλει το Συμβούλιο να θέσει δεσμευτικού στόχου, αν θυμάμαι καλά. 26 υπουργοί ήταν κατά των δεσμευτικών στόχων και ένας μόνος τους ήθελε τους δεσμευτικούς στόχους. Η οδηγία για τα δεσμευτικά μέτρα βρήκε αντιμέτωπη την πλειοψηφία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό και δεν πέρασε κανένα μέτρο. Επομένω, εσεί τι στόχο έχετε θέσει για να πετύχετε το στόχο. Τι θα γίνει δεν καταφέρετε το 20% από ό,τι φαίνεται για την αποτελεσματική χρήση ενέργεια. Τι λέτε. ich habe auch noch zwei, drei kleine Ωραία. Ε? Πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, ε, καταρχά πρέπει να επενδύσουμε σε εργοστάσια. Υπάρχει και αυτή η ανάγκη. Και στη δική μου τη χώρα υπάρχει το πρόβλημα σε... Κάποιοι επενδυτές δεν θέλουν να επενδύσουν σε τέτοια σε περιπτώσεις γιατί λένε ότι ε, ήδη έχουν επενδύσει σε άλλα εργοστάσια και σε άλλα δίκτυα λόγω της εσωτερικής αγοράς. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει πρόβλημα λόγω του τρίτου πακέτου για την εσωτερική αγορά. Υπάρχει περίπτωση να διευκρινιστεί με κάποιο τρόπο αυτό. Δεύτερον, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Είπατε ότι χρειάζεται πιο έντονη έτσι, κοινωνικοποίηση της ε, ε, ενέργειας πώς, για τις ανανεώσιμες πηγές. Πώς ακριβώς το ε, εννοείται αυτό. Δηλαδή θα αντικατασταθούν τα προγράμματα από τα κράτη-μέλη με κάποιο ευρωπαϊκό για να είναι πιο υψηλή η αποτελεσματικότητα. Κλείνει το μικρόφωνο του Πρόεδρου όμως. Τρίτον, Πώς εκτιμάτε τις συνέπειες των ε, αποφάσεων που λαμβάνονται για την ενεργειακή πολιτική ε, από την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Ε, τις τελευταίες εβδομάδες κάνουμε πάρα πολλές συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή ε, Βιομηχανία η οποία όντως επίγεται να έχει συγκεκριμένα μέτρα και αυτή η συζήτηση γίνεται όλο και πιο συχνά και για το πρόβλημα της επιβάρυνσης και του κόστος της ενέργειας. τελικά τα όρια που βρίσκονται για το πώς επιβαρύνουμε και πώς επιβαρύνουμε την, ε, ε, την βιομηχανία με την ενεργειακή μας πολιτική. Γιατί δεν μιλούμε μόνο για τους στόχους για την παραγωγή του, του του άνθρακα, αλλά και το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε, να εξακολουθήσουμε να διατηρούμε τη βιομηχανία στην Ευρώπη. Δεν έχω άλλα ερωτήματα, δεν μου έρχεται και τίποτα άλλο να ρωτήσω, οπότε ο Επίτροπος έχει το λόγο. Πρόεδρε, να ξεκινήσω από το τελευταίο σας ερώτημα. Αν δούμε την κατάσταση του, που υπήρχε τον Νοέμβριο του 2009, το 2011, συγγνώμη, η Ευρώπη, αν τα πάει καλά, θα έχει ε, απόλυτη στασιμότητα αν τα πράγματα πάνε άσχημα και θα έχει απλώς ύφεση αν τα πράγματα πάνε καλά. Έτσι είναι τα πράγματα. Ε, μέχρι την, τον επόμενη χρονιά τουλάχιστον δεν θα έχουμε ανάπτυξη. Θα έχουμε τουλάχιστον 10 κράτη-μέλη με ύφεση και θα έχουμε σε αυτά τα κρατημέλη που κάτι αναπτύσσεται μια οριακή ανάπτυξη. Και γι' αυτό η ευφυής ενεργειακή πολιτική για την οικονομία, για την ε, βιομηχανία θα γίνεται όλο και πιο ευαίσθητη και βεβαίως πιο σημαντική. Φυσικό, φυσικά πρέπει, ας πούμε, κράτη όπως η Ιταλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Τσεχία, να δούμε ε, και το κόστος ε, για την ηλεκτρική ενέργεια αλλά και τις ε, πρώτες ύλε που υπάρχουν. Γιατί αυτά παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από το κόστος των θέσεων εργασίας. Μιλούμε δηλαδή για την χαρτοβιομηχανία, το αλουμίνιο, τα κεραμικά, τρόφιμα. Μιλάμε για πάρα πολλούς, για τη χημική βιομηχανία. Μιλάμε για πάρα πολλούς τομείς που επηρεάζονται. Οπότε εγώ είμαι διαθέσιμος, γιατί εσείς είστε ακριβώς η Επιτροπή για τη βιομηχανία και για την ενέργεια και το θέμα της, ε, της πολιτικής, της περιβαλλοντικής επίσης είναι σημαντικό, να συζητήσω μαζί σας για το ποια πολιτική θα διατηρήσει τις ε, θέσει εργασία και ποια τελικά είναι η πολιτική που θα κινητοποιήσει τη βιομηχανία. Για τα συγκεκριμένα τώρα ερωτήματα. Όταν λέτε ότι δεν θα θέλαμε να κλείσουν τα πυρηνικά εργοστάσια. Όχι, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Ε, σήμερα είμαι ουδέτερος αντικειμενικά. Είπα ότι το stress test ούτε θα αποτελέσει ένα τεστ που θα δώσει τη σφραγίδα για όλα τα ε, πυρηνικά εργοστάσια, ούτε όμως θα δημιουργήσει αυτοματισμό. Συνέπειες τώρα και για την κατάσταση των, εργοστασίων, για την ε, ε, προμήθεια, ε, για το κόστος, για την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, ότι μπορεί κάτι να μην αξίζει τον κόπο πια να λειτουργεί, ας πούμε, οι άλλες προτάσεις που μπορεί να γίνουν, θα σίγουρα θα υπάρξουν. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρξουν όλες αυτές οι συνέπειες. Την έκθεση λοιπόν αυτή δεν μπορούμε να την υποβάλουμε πριν τον Μάρτιο-Απρίλιο του επόμενου έτου. Γιατί? Γιατί κάνουμε ένα stress test σε τρία επίπεδα. Πρώτο επίπεδο, ε, ναι, ε, εξέταση που την έχουμε ήδη κάνει των δικών μα εγκαταστάσεων. Δεύτερη φάση, τα μέσα των ρυθμιστών του τα κράτη-μέλη ελέγχουν. Και, και χρειάζονται ε, χρόνο, για, μέχρι το, τον Δεκέμβρη σίγουρα τα κράτη-μέλη. Και μετά έρχονται οι εκθέσει των κρατών μελών σε εμά. Οπότε, ξεκινούμε με το peer review ε, τον Γενάρη, που σημαίνει ότι οι Αυστριακοί θα ελέγξουν ε, τους, ε, κάποιους στην Γαλλία, οι Φιλανδοί θα ελέγξουν το Βέλγιο, οι Ολλανδοί θα ελέγξουν ε, τους Σλοβαίνους. Θα ξεκινήσουν λοιπόν αυτές οι, αυτά τα τεστ, αυτή η έλεγχη και μετά θα χρειαστούν 8 με 10 εβδομάδες. Και μετά προφανώς θα, θα χρειαστεί να γίνει και μια σύνοψη όλων αυτών. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, μην περιμένετε την έκθεση πριν τον Απρίλιο. Αλλά ε, σίγουρα θα είμαστε ε, πολύ οξυδερικοί σε όλο αυτό, θα κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά, λεπτομερέστατη. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από την ταχύτητα. Επίση, πρέπει να δούμε ποιε θα, είναι οι συνέπειε για την ε, νομοθεσία, την απτή, για να επιτύχουμε μεγαλύτερη πυρηνική ασφάλεια. Έχουμε ε, την ε, εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όχι για το 2014, αλλά ήδη από τώρα να κάνουμε την ανανέωση της οδηγίας για την ε, πυρηνική ασφάλεια. Οπότε ερχόμαστε κατευθείαν στο 2012. Τώρα, για το τρίτο πακέτο της εσωτερικής αγοράς. Πέρσι και στο πρώτο εξάμεινο του 2011 ε, είχαμε κάνει διαβουλεύσεις, είχαμε συμβουλεύσει τα κράτη-μέλη. Το Σεπτέμβριο είχαμε μεγαλύτερο αριθμό, ξεκινήσει μάλλον μεγαλύτερο αριθμό διαδικασιών επί παραβάση. 18 περίπου κράτα οι μέλη που έχουν καθυστερήσει τις διαδικασίες τους και στο αέριο και για την ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά και αυτό είναι το μόνο μα όπλο. Είμαστε ενώπιον του δικαστηρίου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε Κάποια κράτη-μέλη εφάρμοσαν ε, ή θα εφαρμόσουν εθελοντικά το πρόγραμμα αυτό ή θα έρθει η αποφάση του δικαστηρίου εν αυτό το χρόνο και θα χρειαστεί υποχρεωτικά να την εφαρμόσουν. Μετά. Όταν ε, ξεκινούν οι πρώτες ε, διαδικασίες ε, για τους, με τους Ρώσους για, τον, για την Gazprom, ο πρόεδρος Μετβέντεφ έχει πει ότι αν η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν αρκεί, τότε μάλλον θα πρέπει να την αλλάξουν. Δηλαδή τη δική μου αξιολόγηση είπε. Το τρίτο πακέτο ενέργειας θα αρκέσει. Απλώς δεν γίνεται αποδεκτό. Αυτό είναι άλλο. Η Gazprom και οι Ρώσοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι, τα καταλαβαίνουν όλα, αλλά απλώς δεν τους αρέσει, δεν τους συμφέρει. Οι Ρώσοι θέλουν ιδιοκτησία του αερίου, των εταιριών αερίου, των αγωγών, των επιτόπου εργοστασίων και όλων όσων φοράνε τη φανέλα της Γκάσπρομ. Θέλουν δηλαδή ιδιοκτησία όλη της αλυσίδας. Και εντάξει, αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε το 2009. Αλλά εσείς και το, κοινοβούλιο, ε, και το Συμβούλιο συγγνώμη, αποφάσισαν όχι. Οπότε έχουμε διαχωρισμό της μεταφοράς και της παραγωγής. Και αυτό θα τηρήσουμε. Ε, και οι ευρωπαϊκές ε, εταιρείες και οι τρίτες χώρες. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μεταφέρετε αέριο από την Νορβηγία σε εμά. Οι Νορβηγοί δεν παραπονούνται. Ούτε οι Αλγέροι ε, παραπονούνται. Αλλά οι Ρώσοι δεν θέλουν και πιέζουν την κατάσταση. Βεβαίω οι Ρώσοι παραμένουν ο πιο σημαντικό μα τέρο, αλλά η δράση φέρνει αντίδραση. Γι' αυτό το κατάλαβαν οι Ρώσοι και κάποια στιγμή θα πρέπει και να το αποδεχτούν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να του κάνουμε να το δεχτούν. Οπότε, παρά το, τα όσα είπε η ε, Καγκελάριο, το τρίτο πακέτο δεν μπορεί να αλλάξει αν μπορούσε να αλλάξει, θα έπρεπε να υπάρξει πρωτοβουλία της Κομισιόν, που δεν θα την αναλάβουμε εμείς, και χρειάζεται απόφαση του Κοινοβουλίου, το οποίο μάλλον εσεί δεν το θέλετε. Οπότε, όλα τα, όλοι οι είναι στο μανίκι μας. Και για το θέμα του South Stream ο South Stream μέχρι στιγμή έχει, έχει μια χοντρική, έτσι, ένα χοντρικό σχεδιασμό. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη, ακόμα και, τα, και οι χώρε που έχετε εσεί στι εκλογικέ σα περιφέρειες και εν μέρει και κάποιε κυβερνήσει στι οποίε ανήκουν ε, και οι δικοί σα όπαδοι, έχουν δεσμευτεί για τον South Stream, το δέχονται δηλαδή. Αλλά βεβαίω αυτό δεν μα διευκολύνει καθόλου τη ζωή. Δεν υπάρχει ακόμα ε, εξαίρεση, δεν υπάρχει σύμβαση, δεν υπάρχει τίποτα για το τρίτο πακέτο για την ε, ενέργεια. Οπότε μέχρι στιγμής ο South Stream δεν έχει ξεκινήσει, δεν βρίσκεται δηλαδή σε καμιά διαδικασία λήψης απόφασης. Αν ε, ο σχεδιασμός συνεχίσει έτσι όπως έχει και εσείς ε, και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερωθούμε για τις προθέσεις του, των Ρώσων εταίρων μας, έτσι ώστε να μπορούμε μετά να λάβουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά την απόφαση. Αλλά διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποιοι, κάποιες ευρωπαϊκές εταιρείες φυσικού αερίου, μάλιστα μία γερμανική και μία γαλλική, που είναι κρατικές εταιρείες η ΖΕΝΤΕΦ έχει εμπλακεί. Για το σχιστολιθικό αέριο έχουμε σαφή θέση. Αν τα κράτη-μέλη ε, δεχτούν τέτοια project και αν τα κράτη-μέλη θέλουν να τηρήσουν και το ευρωπαϊκό δικαίο για, ε, για, το, ε, για το περιβάλλον και το εθνικό τους δίκαιο, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είμαστε υπέρ. Μάλιστα στην Πολωνία, προς το παρόν, τώρα, ε, υπάρχουν τέτοιε δοκιμές. Νομίζω ότι το ε, σχιστολιτικό αέριο δεν ε, αντικαθιστά το φυσικό αέριο, αλλά είναι ένα, μια, μια προσθήκη, ας πούμε, κάτι επιπλέον στο συμβατό αέριο και στα αποθέματα που υπάρχουν. για τον ορίζοντα 2020 και την ε, έρευνα. Εγώ είμαι σε πολύ καλή επαφή με την Επίτροπο ε, Κεν και όλα τα προγράμματα που έχουμε θα τα προωθήσουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα και επίσης θα λάβουμε από ό,τι φαίνεται και περισσότερα κονδύλια. Ε, στο, η, εφτα, αυτή ε, η, της, δημοσιονομικών να έχει μια προοικοδότηση 80 δι. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια καλή απόφαση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Στο, στη διάσκεψη που έγινε στο Κάβαρα την, προηγούμενη εβδομάδα, όλοι ε, έμειναν με το στόμα ανοιχτό ότι η Ευρώπη ξαφνικά δεν έχει χρήματα λόγω της ε, κρίσης του ευρώ αλλά ότι μπορεί να τηρεί δεσμεύσει και συμβάσεις χωρίς να έχει λεφτά, τους ε, εκπλήσει. Εμεί θέλουμε να έχουμε δυνατότητα διαπραγματεύσεων ε, και ελπίζω το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να βρείτε μια καλή ε, λύση. Από τα 80 δις, ο 10 με 13% θα πάει στην, ενέργεια, στην έρευνα για την ενέργεια. Και όταν ξέρουμε τι έχουμε αναέτος, θα μπορούμε να συζητήσουμε του χρόνου για το ποια θα είναι τα σημεία κλειδιά για την έρευνα και την ενέργεια. Ώστε μέχρι το 2014 να έχουμε κάτι απτό στα χέρια μας. Επίσης υπήρξε το ερώτημα των εξορίξεων offshore. Δεν θέλουμε ύψιστα όρια να καθορίσουμε για την ε, ασφάλεια, θέλουμε ελάχιστα πρότυπα το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε καλό επίπεδο, ας πούμε, στα, για τα πρότυπα που υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν, ας πούμε, οι Νορβηγοί που έχουν δύο-τρία πιο αυστηρά πρότυπα. Δηλαδή, για μας ε, πρέπει να δούμε και το θέμα της, των βέλτιστων πρακτικών. Ας πούμε, στην ε, Μεσόγειο ή στην ε, Μαύρη Θάλασσα υπάρχουν χαμηλότερα πρότυπα. Αλλά κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να θεσπίζει μόνο αυστηρά πρότυπα. Και από πρώτες ε, συζητήσεις που έχουμε κάνει ε, στο Λονδίνο με ε, αξιωματούχους της κυβέρνησης και με πετρελαϊκές εταιρείε, είδα ότι υπάρχει μια ανησυχία, ότι η... υπάρχει και από εμά και από εσάς έτσι, μια προτίμηση για ευρωπαϊκή οδηγία για τον τομέα αυτό. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο κάτι τέτοιο. Μετά, το ερώτημα των ε, προτύπων για την ασφάλεια των ε, πυρηνικών εγκαταστάσεων. Και πάλι πάμε στο Λονδίνο. Το Λονδίνο ναι, ναι. έχει μια πολύ καλή κατανόηση του θέματος της ασφάλειας, αλλά μο, πολύ, ελάχιστη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον τομέα αυτό. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι ευχαρίστως να λάβουμε όποια υποστήριξη γίνεται για να για να δούμε κατά πόσο η Βρετανική ε, κυβέρνηση μπορεί να θέσει τόσο αυστηρά ή αν θα μπορεί να δεχτεί η Βρετανική κυβέρνηση τόσο αυστηρά πρότυπα για, την, για τις εταιρείε της. Οπότε τον επόμενο ε, χρόνο θα έχουμε μία αξιολόγηση επιπτώσεων και θα γίνει και μια πρόταση, για την, ε, πρόταση νομοθετική. Οπότε ε, ο συνάδελφος ο Κλοντ Τιούρμες και άλλοι είναι σε επαφή μαζί μας και την επόμενη χρονιά θα μπορέσουμε να υποβάλουμε και μία πρόταση. Τώρα για το θέμα που ρωτήσατε. Πώς θα μπορέσουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα να προχωρήσουμε. Καταρχάς μιλούμε για τυποποίηση. Έχουμε τα ΕΦΗ e, δίκτυα. Έχουμε την πρότασή μας που θα ψηφιστεί την επόμενη χρονιά. Μετά θα έχουμε μεγάλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, ας πούμε Βορειοδυτική Ευρώπη, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Γερμανία, κάτω χώρες, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Γαλλία, συν τον εταίρο μας την Νορβηγία. για το αέριο και το δίκτυο ηλεκτρισμού της Βορείου Θάλασσας. Και εκεί θα γίνει και μεταξύ αυτών θα γίνει η ε, συζήτηση έτσι ώστε ό,τι αποφασιστεί να αποφασιστεί και να εφαρμοστεί ταυτόχρονα. Επίσης, έχουμε τους ρυθμιστές που θα πρέπει να δούνε το σύστημα των, ε, των, της το κόστος μεταφοράς και θα πρέπει να υπάρχουν συγκρίσιμες τιμές έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν επενδύσεις και από τους ιδιώτες και από τις τράπεζες. Ε, Energiearmut nehmen wir ernst. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι τιμές της ενέργειας να μην αυξηθούν χωρίς να υπάρχει λόγος. Αν αυξηθούν εντάξει, αλκεί όμως να έχουν γίνει επενδύσεις. Αλλά τώρα δεν υπάρχει λόγος να παίζουν ρόλο ε, παράγοντες που να ε, αυξάνουν το κόστος χωρίς να υπάρχει λόγος. Δαπάνες, ας πούμε, ή φόροι σε ε, εθνικό επίπεδο. Το θέμα πρέπει να είναι μια ενέργεια η οποία να μπορεί, την πονήπη να μπορει την να πληρώσουν οι πολίτες. Εμείς για τον άνθρακα και τις εκπομπές διοξιδίου και τον στόχο του 20% είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σύμφωνα με το, τα, και τα κράτη-μέλη και εμείς προχωρούμε σύμφωνα με τα σχέδια που έχουμε. Αν τα επόμενα χρόνια ξεπεράσουμε το στόχο που έχουμε θέσει για, τον, για το διοξείδιο του άνθρακα, αυτό μπορεί να είναι η, ο λόγος μπορεί να είναι η κρίση, η οικονομική κρίση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε την μείωση των εκπομπών ως, και ως καινοτομία. Γιατί όσο πιο πολύ αυξάνεται η κρίση, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να επιτύχουμε το στόχο. Πρώτο τελευταίο σημείο. Θέλουμε νέους δεσμευτικούς στόχους αυτό το θεωρώ πιθανό, αλλά όχι υποχρεωτικό. Ευχαρίστω στα πλαίσια της, και όσο θα εξελίσσεται η συζήτηση για τον ροδικό χάρτη για την ενέργεια, να το συζητήσουμε. Εγώ είχα έναν πιο υψηλό στόχο για την μείωση των, του, των του άνθρακα. αν θέλουμε το 2050 να έχουμε μηδενική, α, μηδενικές εκπομπές του άνθρακα, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 30% μείωση, 30% ε, περισσότερο από ό,τι έχουμε τώρα. 20% στο πρωτογενές ενεργειακό μείγμα και 20% από τον ε, τομέα των μεταφορών, που σημαίνει βιοκαύσιμα για τις μεταφορές. Για τα βιοκαύσιμα Πρώτη γενιάς, εγώ δεν έχω πιστεί ακόμα. Όσο δεν πλησιάζουμε τα βιοκάψιμα δεύτερης γενιάς, και όσο η έλλειψη κινητικότητας αποτελεί πρόβλημα, νομίζω ότι για τη βενζίνη και το ντίζελ για τα αυτοκίνητα και για τις μεταφορές γενικώ, θεωρώ ότι δεν, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα πιο υψηλό στόχο. Οπότε ας δούμε την ε, έρευνα, ας δούμε την κοινοτομία, ας δούμε τους στόχους που έχουμε θέσει και ας ε, φροντίσουμε να τους επιτύχουμε. Τώρα, για το 20% για, την, ε, για το ενεργειακό μείγμα, αν έχουμε ας πούμε στο 10% το, την, τις μεταφορές και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 35%, ως στόχους και, θα, και γίνουν αποδεκτοί ας πούμε από το κρατη Η η Αυστρία μπορεί να ξεπεράσει το 35, να πάει στο 50, η Δανία στο 40, ε, μέσος όρος 35. Ε, Αν έχουμε ε, υψηλότερο δεσμευτικό στόχο για το 2030 και θέλουμε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τέτοιο στόχο πιο ψηλό, ας πούμε 55% στον τομέα του ηλεκτρικού, της ηλεκτρικής ενέργειας, θα χρειάζεται επί τη βάση της ε, ισχύουσας συνθήκης της Λισαβόνας συμφωνία και των 27 κρατών μελών. Αυτό δεν θα περάσει με πλειοψηφία γιατί η αρμοδιότητα έγινε στα κρατημέλη για το ενεργειακό μείγμα. Συμφωνία λοιπόν όλων, ομοφωνία των 27 κρατών μελών. Ας βγάλουμε τις δύο μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Ε, θα συμφωνήσουν ε, οι 25 για το, ε, για το 55%. Η Πολωνία, ας πούμε, που χρησιμοποιεί 90% άνθρακα για, το, για την ενέργεια. Φαντάζεστε οι Πολωνοί να, πάνε, να πρέπει να πάνε στο 55% άνθρακα, χρήσης άνθρακα. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουν. Οπότε, ας μην έχουμε τεράστιες προσδοκίες οι οποίες τελικά γίνονται ψευδεστήσεις. Μετά, η Γαλλία. Έχει 60% πυρηνική ενέργεια, 60-70% πυρηνική ενέργεια. Ε, μπορείτε να φανταστείτε το 2030 να το πάει στο 55%? Μπορεί η Γαλλία ίσω αν την κινητοποιήσουν οι πράσινοι, αλλά δεν νομίζω ότι η Σαρκοζή θα το δεχτεί. Τη συζήτηση λοιπόν αυτή ευχαρίστως να την κάνουμε, γιατί όσο υπάρχει η συνθήκη και είναι έτσι όπως είναι, δεν μπορούμε να θέσουμε πιο υψηλούς ε, στόχους ε, για την ενέργεια και να είναι και δεσμευτική. Μετά, ενεργειακή απόδοση. Εγώ περιμένω ε, ειλικρίνεια. Ο συνάδελφο Μπένσον, όπω και άλλοι, είπαν εδώ ότι θέλετε πιο δεσμευτικού στόχου. 20% και δεσμευτικό ω στόχο. Εγώ ε, έχω συζητήσει πολλέ φορέ με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Θα Μάλιστα, συζητούμε αύριο το πρωί για το θέμα αυτό. Αύριο το πρωί στι 10 συγκεκριμένα. Το Συμβούλιο το αρνείται με μεγάλη πλειοψηφία. Ίσως η Δανία να δεχτεί. Αλλά το Συμβούλιο με τη, στη μεγάλη του πλειοψηφία το αρνείται. Το απορρίπτει. Οπότε δεν έχει νόημα να οδηγούμε προς έναν τοίχο. Τώρα, οπότε έχουμε μέτρα τώρα και σε δύο-τρία χρόνια, αν τα μέτρα δεν λειτουργήσουν, τότε δεσμευτικούς στόχους. Αλλά να έχουμε τώρα ε, μία έτσι ε, πανάκια για όλα δεν, δεν γίνεται. Γι' αυτό έχουμε το 1,5% ε, μείωση αναχώρα ή ανα εταιρεία. Γι' αυτό έχουμε το 3% για τα δημόσια κτίρια. Και τώρα τα κρατημέλη κάνουν και αυτά πίσω και λένε χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία. Εγώ ευχαρίστω. Είμαι υπέρ τη ευελιξία. Τα κράτη-μέλη μπορούν να, ε, μπορούν να έχουν, ε, ε, δεν μπορούν να έχουν και τα δύο, όχι ούτε μέτρα, ούτε δεσμευτικούς στόχους και ευελιξία και να επιτύχουμε τον ελάχιστο, ε, τον, τους ελάχιστους στόχους. Δεν γίνεται. Στο κοινοβούλιο θα έλεγα ότι είναι. Υπάρχουν διάφορες ε, απόψεις. Αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να συμφωνήσουμε. Στο Συμβούλιο όμως αυτό ε, υπάρχει τεράστια διαφορά ακόμα και από τη μία μέρα στην άλλη. Κάθε Κυριακή ε, λένε ότι περιμένουμε το, το, το κατώτερο δυνατό. Η ε, ενεργειακή απόδοση είναι η πιο φτηνή ενεργειακή πηγή, ε, τη μία μέρα, την άλλη μέρα λένε το εντελώ αντίθετο. Α πούμε, πάρετε ένα νοσοκομείο ή ένα, ένα κτίριο και θέλουμε, που θέλουμε να το κάνουμε ενεργειακό αποδοτικό. Από, από, από την ταράτσα του μέχρι, την, ε, μέχρι το, τους ε, καυστήρες του. Το οποίο θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο χρόνια για να αποσβέσει τα χρήματά του. Η γενιά άνω των 60 είναι α, διατεθειμένη να επενδύσει. τα παιδιά τους όμως, η αμέσως επόμενη γενιά, δεν συμφωνεί. Bei der Politik, die sagen, alle haben kein Geld, die Krise. Οι πολιτικοί λένε δεν έχουμε λεφτά, μειώνονται οι προϋπολογισμοί μας, έχουμε κρίση και στο Βερολίνο, μην νομίζετε, και στη Στουτγκάρδη. Αλλά και στην Αθήνα και στη Μαδρίτη και στη Λισαβόνα και στο, Λουβδί, και στο Δουβλίνο και αλλού. Η ενεργειακή απόδοση ε, συνήθως ε, την παραβλέπουμε λόγω των ε, οικονομικών προβλημάτων. Και οι επενδύσεις στον τομέα αυτό θα επιτύχουν μόνο αν, αν θεωρηθεί προτεραιότητα ενεργειακή απόδοση. Οπότε μετά θα πρέπει να δούμε αν το σχολείο θα πρέπει να είναι ενεργειακό αποδοτικό, ενεργειακός αποδοτικό, ε, αλλά θα πρέπει να έχει περισσότερα παιδιά σε κάθε τάξη γιατί θα υπάρχουν λιγότεροι δάσκαλοι. Ε, εκεί καταλήγει η συζήτηση. Ή θα πρέπει να έχουμε λιγότερου αστυνομικού, αλλά μία, ε, ένα ενεργειακό αυτόνομο και αποδοτικό εκτίριο για την αστυνομία. Είμαστε λοιπόν σε μια πολύ έντονη συζήτηση και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μόνο οι επενδύσεις είναι αυτές που θα βοηθήσουν, παρόλο που μετά από δύο δεκαετίες θα ε, αποσβεστούν τα χρήματα των επενδύσεων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Εγώ ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο επόμενος ε, Επίτροπος είναι ήδη εδώ.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 Dámy a pánové, budeme pokračovat v podstatě v tématu θα ασχοληθούμε με τα θέματα ενέργειας και θα ήθελα να ρωτήσω, να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί ο πρόεδρός μας μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Επομένως από εδώ και πέρα τσεχικά θα ακούτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο, τον κύριο Ποτόσνικ, ο οποίος ε, ήρθε εδώ για να μας παρουσιάσει πολύ σημαντικά θέματα. για την αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων και για να μην καθυστερούμε, να μην χρονοτριβούμε, θα, έχει μια παρουσίαση, θα κάνει μια παρουσίαση ο Επίτροπος 15 λεπτών περίπου και μετά θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, μέλη της, αγαπητά μέλη της Επιτροπής. Καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ ωραίο που είμαι ξανά στην παλιά μου επιτροπή. Είχα τακτικές επαφές με την Ήτρε όταν ήμουν επίτροπος για τις επιστήμες ε, και την έρευνα. Και ήθελα πάρα πολύ να έρθω εδώ και να σας εξηγήσω και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της, ε, του περιβάλλοντος. Γιατί, διότι τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούσα να τοποθετήσω ε, την ε, περιβαλλοντική πολιτική στους οικονομικούς, βιομηχανικούς και ε, τομείς ε, πολιτικής και στην πολιτική καινοτομία. Νομίζω ότι το περιβαλλοντικό, η περιβαλλοντική νομοθεσία η οποία πέρασε από το, κοινοβούλιο, από το σας προσφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες ένα πιο καθαρό αέρα και νερό, τιμωρεί τους, ε, αυτούς που μολύνουν και θα πρέπει να ε, συνεχίσει να ε, υλοποιεί αυτούς τους στόχους. Είναι πολύ καλύτερα, αλλά είναι πάρα πολύ καλύτερα να προσφέρουμε τα μέσα και τα κίνητρα για να είμαστε σίγουροι ότι δεν μολύνουμε ευθύ εξ αρχή ε, και ότι η συμπεριφορά μας και η παραγωγή μας και η κατανάλωσή μας είναι βιώσιμες μέσω του κύκλου ζωής των προϊόντων και ε, καθ' όλη τη διάρκεια της αλυσίδας προμηθειών. Ας δούμε ποια είναι η ποιες πώς τοποθετείται τώρα η συνολική μας ανταγωνιστικότητα που συνδέεται με την ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικό τους πόρους. Α δούμε καλύτερα. Κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα ο πληθυσμός ε, της, ε, του πλανήτη μας τετραπλασιάστηκε και η οικονομική μας παραγωγή τε, τε, ε, πολλαπλασιάστηκε 40 φορές. Έχουμε αυξήσει τα ορυκτά μας καύσιμα 16 φορές, χρησιμοποίησαμε 16 δηλαδή φορές περισσότερα ε, ορυκτά καύσιμα, τα αλλιεύματα μας αυξήθηκαν κατά 35 φορές και έχουμε χρησιμοποιήσει 9 φορές παραπάνω ε, το, το νερό που είχαμε στη διάθεσή μας. Αυτό λέγεται μεγάλη επιτάχυνση. Με έναν παγκόσμιο πληθυσμό 1,5 δισεκατομμύρια πριν από 100 χρόνια, αυτή, το, μονοπάτι, το μονοπάτι ανάπτυξης ήταν εντάξει. Μας έδινε υγεία, ευημερία και υγεία. Όμως ε, ε, το, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι έχουμε ένα πληθυσμό 7 έως 9 δισεκατομμύρια. Επομένως το μονοπάτι αυτό δεν είναι πλέον βιώσιμο. Επομένως το business as usual, το οποίο ήταν ένα σενάριο ε, που θα μπορούσε να ισχύσει πριν από λίγα χρόνια, τώρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι δεν θα έχουμε πλέον πόρους, τους απαραίτητους πόρους μέχρι το 2050. Επομένως το πρώτο μου μήνυμα είναι ότι η αποτελεσματικότητα των πόρων δεν είναι είναι μια επιλογή, είναι ε, κάτι το αναπόφευκτο. Και η επιλογή μας δεν είναι αν θα αναπτύξουμε, αν θα αναπτύξουμε τώρα ή κατά πόσο θα περιμένουμε μέχρι όταν αναγκαστούμε ε, όταν πλέον οι κρίσιμοι πόροι έχουν ε, εξαφανιστεί ή είναι πλέον ιδιαίτερα δαπανηροί. Η θέση της Ευρώπης όσον αφορά την, την ανέβρεση των πόρων που έχουν γίνει πλέον δυσέβρετη δεν φαίνεται και τόσο καλή. Όπως ε, ε, είπατε και στην έκθεση του κύριου Κόφερ, είμαστε φτωχοί όσον αφορά τους ορυκτούς, ε, τους ορυκτούς πόρους. Έχουμε το, παίρνουμε το 48% του χαλκού των κοιτασμάτων χαλκών από το εξωτερικό, το 64% του ψεδάρου και του βοξίτη και το 78% του, του νικελίου. Επίσης εισάγουμε όλη, όλη, όλες ποσότητες που χρειαζόμαστε για το κοβάλτιο, το, την, ε, την πλατίνα, το τιτάνιουμ και το βανάδιουμ. Είμαστε επομένω μια ήπειρο η οποία εξαρτάται πολύ από τι εισαγωγέ. Ε, ο λόγος, ε, ε, επομένως, πρέπει να, να χρησιμοποιούμε με ικανοποιητικό τρόπο και αποτελεσματικό τρόπο τους πόρους μας. Ο λόγος τον οποίο δεν το κάνουμε είναι γιατί οι τιμές, οι τιμές τους μειώνονταν σε πραγματικούς όρους τα τελευταία 150 χρόνια. Εκτός ε, από τις ε, ε, περιόδους των πολέμων και των πετρελαϊκών κρίσεων. Ταυτόχρονα η τιμή της εργασίας αυξήθηκε. Για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί πρέπει να χρησιμοποιούμε όλοι μας την ευφυΐα για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε αυτά το, αυτό το αυξημένο κόστος με τις ε, σημαντικές αυξήσεις στην ε, παραγωγικότητα της εργασίας αλλά οι μέρες όμως των φτηνών και άπειρων πόρων έχουν τελειώσει. Οι τιμές των πρώτων υλών αυξάνονται τα τελευταία, την τελευταία δεκαετία και έχουν εξαφανίσει τελείως τις μειώσεις που είχαμε τον προηγούμενο, τον προηγούμενο αιώνα. Είμαι σίγουρος ότι το αόρατο χέρι των, ε, που αυξάνει τις τιμές των πρώτων υλών θα κάνει, θα κάνει κάποια από τη δουλειά που πρέπει να γίνει έτσι ώστε τελικά να προσανατολιστούμε προς την αποτελεσματικότητα των, των πόρων. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι τιμές δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την, την έλλειψη ή τις συνέπειες στο περιβάλλον μια σωστά λειτουργούσα αγορά δεν υπάρχει για τον καθαρό αέρα, για τον καθαρό νερό, για τα ψάρια, για τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος εν γέννη. Είναι δικό μας ε, καθήκονο σαν ε, νομοθέτες και καθορίζονται την πολιτική να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι κρίσιμες και ευαίσθητες, ευαίσθητοι πόροι ε, να, ε, πρέπει να, αξιολογούνται και να προστατεύονται και να βοηθήσουμε την βιομηχανία και τους καταναλωτές να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν αυτή την απαραίτητη μετάβαση προσφέροντας τις ε, κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας. Εάν θα πρέπει να αυξήσουμε ε, την ανάπτυξή μας ε, με την καλύτερη χρήση των πόρων, τότε θα πρέπει να δώσουμε σαφή μηνύματα στον επιχειρηματικό κόσμο. Οι Ιάπωνες, οι Κορεάτες, οι Κινέζοι ήδη το έχουν, καταλάβει τι πρέπει να κάνουν. Και αυτό φαίνεται και από τις βιομηχανικές τους πολιτικές. Η πρόκληση για την Ευρώπη είναι ότι μετά από μερικούς αιώνες ε, όπου είχαμε ανάπτυξη εντατική όσον αφορά τους πόρους, ε, κάπου έχουμε μπλοκάρει σε, ε, μέσα, στα, μέσα σε ε, αναποτελεσματικές υποδομές, μέσα σε αναποτελεσματική οικονομική και δημοσιονομική εκμετάλλευση των πόρων. Και το πρόβλημά μας είναι ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε πιο ε, ευέλικτα και έξυπνα προϊόντα, τα οποία να χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους και πρέπει να μπορούμε να πουλάμε ε, αυτές τις συνδυασμένες ε, υπηρεσίες. Επίσης θα πρέπει να αναπτύξουμε και τα οικονομικά εργαλεία έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα δημιουργηθούν, δεν συμβεί σημεία Μέχρι τώρα μίλησα για το τι και για το γιατί. Και από ό,τι κατάλαβα από την γνωμοδότησή σας για την αποτελεσματικότητα των πόρων, ότι το επιχείρημα αυτό το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Ας δούμε τώρα το πώς. Πώς ε, θα ξεπεράσουμε ε, τα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν ε, και να καταλήξουμε σε, σε μια βιώσιμη οικονομία. Ε, πώς μπορούμε να μοχλεύσουμε τις ε, καινούργιες καινοτομίες και ε, έτσι ώστε να κάνουμε τις πρόοδους που απαιτούνται σε κάποιους τομείς. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε τον ε, ιδιωτικό, την ιδιωτική και την δημόσια ζήτηση για τα πράσινα προϊόντα. Αυτό το Αυτά χάρτη... προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε αυτόν τον χάρτη πορείας για τις, τους πόρους της αποτελεσματικής Ευρώπης κλπ. Δεν είναι δικό μου αυτό προσωπικό, είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό εγκρίθηκε από το σώμα των Επιτρόπων και είπαμε έχουμε στο 2050 και πώς να θα Και αυτό είναι, είναι στην καρδιά της ευρωπαϊκή στρατηγικής για ούτω ώστε να έχουμε μια οικονομική μεταρρύθμιση. Και αυτό ήταν η σημαία μας για το 2020, ε, το βασικό μας εργαλείο και αυτό έχει αναγνωριστεί όχι μόνο σαν θέμα του περιβάλλοντος αλλά σαν ε, η ατζέντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη ε, και έτσι λοιπόν με αυτό το θεμέλιο χαρτισπόριας μας οδήγησε σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους. Αυτό είναι το όραμά μας, τόσο να μπορούμε να πετύχουμε ανάπτυξη, να πετύχουμε καλύτερο επίπεδο, όχι σε βάση του περιβάλλοντος και γι' αυτό χρειάζονται κάποιες πρωτοβουλίες απτές. Και ελπίζουμε ότι αυτά όλα τα ορόσημα θα τα έχουμε περάσει η υλοποίηση του 2020 και γι' αυτό θα εστιάσουμε που εκεί που μένουμε σε το τι τρώμε και πώς μετακινούμεθα και για τον απλό λόγο ότι αυτά τα τρία θέματα είναι το 80% των επιπτώσεων των όσων κάνουμε επί τη χρήση των πηγών. Και αυτό ο χάρτη πορεία έχει να κάνει με πάρα πολλά υπάρχοντα εργαλεία πολιτική και όσον αφορά την νομοθεσία για τα απόβλητα μέχρι του διαγωνισμούς, για περιοδικά προγράμματα μέχρι οικολογικά σήματα, αλλά για πρώτη φορά όλα αυτά μπαίνουν σε ένα συνεκτικό λογικό πλαίσιο και έτσι θέλουμε να έχουμε μια τέτοια πολιτική, ε, να έχουμε τέτοιε αποφάσεις για τις επιχειρήσει μέσα στο, στο, στο ευρύτερο οικονομικό μας πρόγραμμα και βέβαια ο χαρτής πορείας δεν λέει όλε τι λεπτομέρειε. Είναι 24 σελίδε και έχει τι νομοθετικέ προτάσει και τι ε, πρωτοβουλίε και επίση έτσι προβλέπονται εκεί πέρα το ποιε είναι, ποια είναι τα ορόσημα, για το 2020, για τις ε, πολιτικοί, ε, οι προτεραιότητες, ε, το τι θα γίνει με τις χωματές του 2020, πώς πρόκειται να καταργηθούν όλες οι βλαβερές επιδοτήσεις μέχρι το 2020, βαθμιαία και για το πώς θα υπάρξει κάποιο είδους περιβαλλοντική φορολογία. Και επίσης για αυτό το λόγο θέλουμε να έχουμε βιώσιμη πολιτική για τα κτίρια, για τα τρόφιμα, χρήση της γης. Αυτά είναι πρωτόγνωρα και για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά το οποίο είπαμε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτές τις επιδοτήσεις. Τα κράτη-μέλη εκταμείευσαν 20 δι όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα για τι σχετικέ μάλλον επιδοτήσεις πέρυσι. Και επίση υπήρχαν κάποιε φορολογικέ ελαφρύνσει για τα εταιρικά αυτοκίνητα που επιβάλλαν 54 δι ετησίω τα 18 κράτη-μέλη, δηλαδή 0,5% του ΑΕΠ αυτή η φύρα ήταν τζάμπα και κακή για το περιβάλλον. Και γι' αυτό τώρα πρέπει να μετακυλήσουμε αυτό το, το βάρος της νομοθεσίας από την εργασία ή στις, στους πόρους ή ε, μόλυνση. Αν θέλουμε να κάνουμε μια τέτοια στροφή θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με τα άριστα των κρατών μελών. Και εκεί θα πρέπει να δούμε ότι έχουμε 1,4% ε, ΑΕΠ όσον αφορά το επιπλέον ε, έσοδο από τους φόρους το οποίο θα μπορούσε αφού εισπραχθεί να οδηγήσει σε συρρήγνωση των άλλων φόρων επί της εργασίας ή να εξυπηρετήσει τα ελλείμματα. Και επομένω με αυτού του δύο τομεί δημιουργούμε τεράστιε ευκαιρίε όσον αφορά κάποιο είδου στέρεα φορολογική πολιτική και γι' αυτό θα δείτε όλοι αυτοί οι στόχοι να εντάσσονται πλήρω ει την ενιαία στατική ανάπτυξη του 2012. Αυτά τα οποία πριν από ε, Λίγε ώρε πριν συζητήσαμε και ε, ε, ταυτόχρονα και τα νοικοκυριά αλλά και η βιομηχανία πρόκειται να έχουν, να έχουν κίνητρα ώστε να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά του πόρου. Επίση με το χάρτη μπορεί να γνωρίζουμε ότι χρειάζονται κάποια όργανα, κάποια, κάποια μέσα πολιτική και για τη ζήτηση και για την προσφορά. Και προ τι δύο κατευθύνσει. Η ιδιαίτερα της προσφοράς θα πρέπει να έχουμε περισσότερη προσοχή στην παραγωγή. Οικολογικό σήμα. Ευρύτερα κριτήρια και όσον αφορά τη ζήτηση να έχουμε μια απλούστερη, ευρύτερη, πιο προσβάσιμη αγορά όσον αφορά τα αηφόρα, βιώσιμα προϊόντα και επίσης να ευθυγραμμίσουμε και να συντονίσουμε το eco-label, το οικολογικό σήμα, το ενεργειακό σήμα και τα κριτήρια για τις, τους πράσινους διαγωνισμούς και προμήθειες του δημοσίου. Κυρίε και κύριοι, είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε κάποιο αξιόπιτη ε, πληροφορία για όλα αυτά. Θα πρέπει να έχουμε ε, τέτοια κίνητρα για την ε, παραγωγή, δεν θα πρέπει να, να, να πριτανεύει ο κινησμό για το θέμα του περιβάλλοντος, θα πρέπει να επιστρατεύσουμε το καλύτερα τους καλύτερους και γι' αυτό το λόγο ε, και οι πολιτικέ μα θα πρέπει να κατατείνουν προ αυτό. Η διαπτωματική χρήση τη ενέργεια θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του τη πολιτική μα. 2012 θα είναι η επόμενη φάση. Σε στενή συνεργασία θα προχωρήσουμε με τον κύριο Ταγιάννη και όλους τους Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, την ε, πραγματική ιδιοκτησία και λίγο και με συνεργασία με τον κύριο Τσόλο. Οπότε, σε τρεις εβδομάδες θα περάσουμε αναμορφησία. Και έτσι θα αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα για την οικολογική καινοτομία όπως την, τεχνολογική ε, γνώση των, των, των επενδυτών να σπάψουν τα ελλείμματα και έτσι να έχουμε καλύτερη περιβαλλοντική έρευνα να εξασφαλίσουμε το ότι οι εταιρείε στην Ευρώπη να είναι πιο αποδοτικές πάνω από 30% έχουμε το κομμάτι που όσον αφορά τη διαχείριση των ε, απορριμμάτων. Όλοι αυτοί οι τομεί αναπτύσσονται 5% ετησίω και θα τριπλασιαστεί αυτή η ανάπτυξη μέχρι το 2030. Όμω, οι μέχρι τη ενέργεια δεν είναι μόνο η η Νομίζω ότι σα έχω πείσει ότι έτσι θέλουμε όλη μας η οικονομία να γίνει πιο αηφόρα, πιο βιώσιμη, πιο ανταγωνιστική. Αύριο ο Μακίντζη πρόκειται να δημοσιεύσει, να δημοσιεύσει αυτή η εταιρεία μια έκθεση ότι η παραγωγικότητα θα αποδώσει 2,8 έως 3,53 μέχρι το 2030 και αυτά τα μέτρα πρόκειται να καλύψουν το 1 τρίτο των πηγών μας. Πάμε. Για 1% μείωση χρήσης πόρων ενεργειακών που θα σε 23 δις ετησίως για τις επιχειρήσεις και 150.000 θέσεις εργασίας και όλοι έχουν καταλάβει μόνος πόσο ωφελεί αυτή η ενεργειακή αποδοτικότητα. Όμως, όμως, έτσι οι εταιρείε βγαίνουν κερδισμένε. Θα περάσουμε και κάποια μεταβατική περίοδο βέβαια. Όλε οι εταιρείε χρειάζονται υποστήριξη. Και εν κατακλείδη, κυρίε και κύριοι, θα πρέπει να αρχίσουμε να διαπιστώνουμε το ότι η, η περιβαλλοντική πολιτική δεν είναι φραγμός. Είναι εξασφάλιση για την ανταγωνιστικότητα. χρησιμοποιούμε τι επιχειρήσει για να προστατεύουμε το περιβάλλον. Άρα, να η ευκαιρία. Έτσι, ορμενώσουμε τι δυνάμει μα. Και το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ήτρε, όπω και η Ένβη, τροπέ Όλα αυτά προ όφελο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Είμαι πεπισμένο ότι το πρόγραμμα για την ε, υπερημερία. Αυτό για τα χρέη, ότι πρόκειται να πάρει το δρόμο του. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις βασικές παγκόσμιες τάσεις, οι πιο σπουδαίες, εκ των οποίων είναι η σπάνης των φόρων, η αλληλεξάρτηση και η συνακόλουθη ε, αδυναμία της Ευρώπης. Οπότε, προσέχετε μην κάνουμε λάθη. Λάθη. Και το μεγαλύτερο λάθος θα είναι να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Commissar. Uh, and uh, in this time for question Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, λοιπόν. Η κυρία Χιούμπνερ είναι η πρώτη. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την παρουσίαση. Μας δώσατε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες ε, πληροφορίες. Χρειαζόμαστε, χρησιμοποιούμε, είπατε, κατά 50% εξωτερικές πηγές. Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για τις ανα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μιλάμε για την ηλιακή ενέργεια, ε, για την αιωλική. Λίγα όμως λέμε για την ε, ενέργεια του, νερού στην Ευρώπη. Σε πολλές, ε, σε, πολλές, κάποιες περιοχές μπορούμε να έχουμε κάποιους, κάποιες λεκάνες ώστε να διατηρούμε το επιπλέον είδωρ και θα μπορούσαμε ίσως να το χρησιμοποιήσουμε και σαν πηγή ενέργειας. Η δική σας η, ε, άποψη για την ανακύκλωση ποια είναι. Θα πρέπει να ανακυκλώνουμε μόνο τα επιπλέον και να ξαναμπαίνουν μετά ανακυκλωμένα, όσα ανακυκλωμένα νέα προϊόντα στην αγορά ή θα πρέπει να πάμε και στις α, χωματερές. Έχουμε πολλές χωματερές σε πολλά κράτη-μέλη και θα μπορούσαμε ίσως όντως να, τα χρησιμοποιήσουμε, να τις χρησιμοποιήσουμε ως τη γη πρώτων υλών. Ε, βέβαια, ίσως ε, να ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και κάποιες εσωτερικές πηγές, όπως είπατε και εσείς στην ε, παρουσίασή σας. Επίσης, η ανακύκλωση θα μπορούσε να περιλαμβάνει όντως και κάποια πτυχή καινοτομία. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει νέε θέσεις εργασίας. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε λύσει 40 ετών. Έχουμε νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις ε, εσωτερικές, στις δικές μας πηγές και να τις χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά. ίσως να πρέπει να χρησιμοποιούμε πηγές που όντως είναι ανακυκλώσιμες και να δούμε την εσωτερική μας αγορά ως πηγή παροχής ε, πόρων για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση που άκουσα. Είμαι τυχερός γιατί είμαι ε, και σχετικά καινούριο μέλος ε, πήρα τη θέση της συναδέλφου μου η οποία έγινε υπουργό στην, ε, στη χώρα μου έχω παρακολουθήσει από πολύ κοντά τα θέματα περιβάλλοντος και βιομηχανίας και προφανώς θα πρέπει η πολιτική που εφαρμόζουμε να μην αποτελεί ένα εμπόδιο για τις ε, βιομηχανίες μας, για τις επιχειρήσεις μας. Ίσα ίσα θα πρέπει η πολιτική να αποτελεί ε, την, ε, την προϋπόθεση για μια βιώσιμη ανάπτυξη του βιομηχανικού κλάδου. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Γιατί ε, όντως ε, ε, υπάρχει και αυτή η εξάρτηση από τις εισαγωγικές όσον αφορά τις ε, πρώτες ύλες στην Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τους ευρωπαϊκούς πόρους, να γίνει περαιτέρω έρευνα για τα, τον ορυκτό, στον ορυκτό πλούτο, να υποφεληθούμε από τα βάση μας. μπορούμε να αναπτύξουμε νομίζω και να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους γιατί είναι ένα ουσιαστικό μέρος μιας βιομηχανικής ανάπτυξης και στη χώρα μου και στις χώρες της Σκανδιναβίας βλέπετε ε, ποιος είναι ο ανταγωνισμός ε, για την ε, καλύτερη χρήση των πρώτων υλών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση όσο το περισσότερο, διότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή περιβαλλοντική πολιτική, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να δούμε και την δική μας εθνική πολιτική όσον αφορά την αξιολόγηση των πόρων. Ευχαριστώ. Δεν ε, κατάλαβα ένα πράγμα, κυρία Επίτροπε. Είπατε για έναν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του κόστους παραγωγής και τιμών. Ε, η εργασία είναι 20% και τα, η πρόταση είναι 40% είπατε. Και εμείς θέλουμε, από ό,τι κατάλαβα, να μειώσουμε όσο δυνατόν το κόστος εργασίας και να αυξήσουμε το κόστος των υλικών για να διατηρήσουμε παράλλαχτες τις τιμές. Γιατί αν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, δεν μπορούμε να έχουμε τόσο, δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να έχουμε ανταγωνιστικό κόστος εργασίας παρά μόνο να το μειώσουμε. Βεβαίως αυτό σημαίνει μείωση μισθών, μείωση συντάξεων, μείωση εισφορών. Ε, ποιος είναι ο ε, μηχανισμός αυτός Ο εργοδότης δηλαδή θα διατηρήσει ή θα, θα εισφέρει αυτές τις εισφορές που είναι η δική του αρμοδιότητα να εισφέρει σε μεταγενέστερη φάση της παραγωγής και θα έχουμε εντατικά τέτοια ε, ε, προϊόντα εντατικής ε, προσπάθειας. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Δεν μπορούμε να έχουμε πόρους ή υλικά, πρώτες ύλες, εάν δεν δαπανίσουμε ενέργεια για να τα εξορίξουμε από τη γη. Μόνο γεωλογική αξία έχουν ε, εάν βρίσκονται μέσα στο έδαφος. Ενώ αν τα χρησιμοποιήσουμε μέσω της χρήσης ενέργειας θα αυξηθεί και η τιμή. Έχουμε και υλικά που ε, έντασης ενέργειας και υλικά που δεν χρειάζονται τόση ενέργεια. Βέβαια θα μπορούσε ίσως η Κομισιόν να μας παρουσιάσει και ένα πίνακα ε, πόρων και πρώτων υλών καθώς επίσης και με το ισοδύναμο της ενέργειας για να δούμε κατά πόσο η τιμή μπορεί να αποτελέσει και τομέα ένταση τη ε, ε, ενέργεια. Ο κύριο Κέλλη έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς ζητάω συγγνώμη γιατί... Επειδή έπρεπε να πάω σε μια άλλη ακρόαση, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω όσα είπατε. Πάντως αυτά που, τα, που άκουσα με εντυπωσίασαν. Ε, κυρίως αυτά όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις επιχειρήσεις για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και όχι το ανάποδο. Ούτω ή άλλω η αλλως η χάνει ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Στην Ευρώπη έχουμε στόχου. 20% μείωση του διοξίδιου του άνθρακα μέχρι το 2020, ίσως και 30%. Κάλλοι λένε ότι θα έπρεπε να είχαμε φτάσει στο 40% μπορούμε να σεβαστούμε αυτούς τους στόχους και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί ή να αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητά μας όταν ε, ο υπόλοιπος κόσμος, οι μεγάλοι παίκτες, είπα, Κίνα, Ιαπωνία, αποφασίσουν ότι δεν θα, πρέπει να, δεν θα ακολουθήσουν τον δρόμο το δικό μας. Και μετά από 5-10 χρόνια τι θα γίνει, εάν εμείς είμαστε καλοί πολίτες που μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, που σεβόμαστε τους στόχους, τους ξεπερνάμε τους στόχους, αλλά οικονομικά τι θα είναι, θα είμαστε σε καλύτερη θέση ή θα είμαστε σε, πιο, σε, χειρότερη θέση. Next, Madame Tikau. Η κυρία Τικάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιτροπό για την παρουσίασή του και θα ήθελα... Και θα ήθελα να αναφερθώ στην βιομηχανία εξόριξης του άνθρακα. Ξέρουμε ότι ο άνθρακας είναι χρήσιμος για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στην πολιτική που πρέπει να ακολουθήσετε στο μέλλον θα πρέπει να, πρέπει να βρεθούν νέες μέθοδοι εξόριξης του άνθρακα που, θα είναι, ε, που δεν θα μολύνουν τόσο το περιβάλλον. Υπάρχουν άλλες χώρες, όπως η Κίνα παραδείγματος χάρη, που έχουν ε, ε, θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία δεν μολύνουν τόσο το περιβάλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε και άλλους πόρους, πόρους που μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε στην Ευρώπη και πόρους που ε, μπορούμε να εξάγουμε χωρίς να μολύνουμε το περιβάλλον. Αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα, όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί ένα κομμάτι του ενεργειακού μείγματος της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Μιλάμε για πρώτες ύλες που ούτως ή άλλως μας λείπουν, το ουράνιο. Η πυρηνική ενέργεια μπορούν, μπορού μπορει με τη σειρά της να μας βοηθήσει να περιορίσουμε τις εκπομπές ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα αυτή να πάρουν μια απόφαση για το ενεργειακό μείγμα. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την αποτελεσματικότητα των πόρων. Βέβαια, η, προφανώς οι πυρηνικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ασφαλείς. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τελείως την πυρηνική ενέργεια. Τώρα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυστυχώς ε, υπάρχουν διάφορα, ε, διάφορα αεολικά πάρκα, διάφορα πάρκα ε, φωτοβολταϊκών τα οποία έχουν κλείσει διότι γιατί, γιατί έχουν κλείσει γιατί το ηλεκτρικό δίκτυο δεν μπορεί να υποδεχθεί όλη αυτή την ενέργεια που παράγεται και μιλάμε για πολλά χρήματα. 5 δισεκατομμύρια στην Ισπανία, 2 δισεκατομμύρια στην, στην Ιταλία. Και όμως πολλά από αυτά τα πάρκα κλείσανε διότι το υπάρχον δίκτυο δεν μπορεί να, να, να, να, να υποδεχθεί αυτή την παραγωγή ενέργειας. Αυτή την ενέργεια που παράγεται. Ένα τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι το πόσιμο νερό το πόσιμο νερό έχει γίνει ένα προϊόν ελληματικό και στην Ευρώπη λόγω ακριβώς των κλιματικών αλλαγών. Ε, υπάρχουν ολοένα και περισσότερες περιοχές που πάσχουν από λειψιδρία. Χρειαζόμαστε νερό και για, τις, για τη γεωργία και για τους πολίτες μας ε, και για τη βιομηχανία πιστεύω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική που να ε, εστιάζεται στην αποτελεσματική χρήση του νερού. Και χρειάζεται προφανώς να γίνουν ε, επενδύσεις και στην έρευνα. Έρευνα για νέα υλικά, νέες μεθόδους. Ευχαριστώ. komisaři, to dotazy mých ε, λοιπόν, Πολλά τα ερωτήματα κύριε Επίτροπε. Να σας δώσουμε το λόγο, να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε όλα αυτά, γιατί είναι όντως πολύ σημαντικά. Παρακαλώ. I will start with uh, Κύριε Χίπνερ, να ξεκινήσουμε όσον αφορά τις ερωτήσεις που μου έθεσε. Βεβαίως. Και το νερό. Α, γιατί ε, για το νερό καλύπτει και την ε, ε, τελευταία, η κυρία Τικάου. Ε, το νερό και η σπάνιση ε, βεβαίω. Το νερό είναι ένας από τους πόρους που τους έχουμε σαν προτεραιότητα. Βεβαίω και έχουμε την οδηγία για τα τα είδη που είναι οδηγία πλαίσιο και εκεί ορίζεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ετοιμάσουν μια τιμολογιακή πολιτική για το νερό. Δηλαδή αντιμετωπίζεται αυτό και σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά επομένως υπάρχει ήδη νομοθεσία σχετική. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να εστιαστούμε για τις δραστηριότητε μας σε κάποιο από τα θέματα που σχέση με τη φύση. Βιοπικιλότητα πέρσι, φέτος αποτελεσματικότητα για την ενέργεια και του χρόνου νερό. Άρα, εργαζόμαστε εντατικά πάνω σε αυτό. Άρα, θα έχουμε ένα σχέδιο για την ε, ασφαλή χρήση των υδάτων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση επί τη βάση των αναλύσεων των όσων θα μας πούν τα κράτη-μέλη σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτων και την κύρια των ποταμών κλπ. Γιατί έτσι κι βέβαια το, το, το, ο εντροφό είναι κοινό στην Ευρώπη. Να δούμε τι γίνεται και με τις ξηρασίες όμως. Και πώς είναι, Βίλιαμ, πώς ήταν το άλλο, το άλλο, α, το άλλο είναι οι πλημμύρες. Έχουμε και το θέμα τη κλιματική αλλαγής. Επομένως, όλα αυτά έχουν αρχίσει να μας απασχολούν και βέβαια η προσοχή μας είναι αμέριστη προς τα εκεί. Και η ανακύκλωση. Επίσης μας απασχολεί. Έχουμε την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Έχει προχωρήσει, έχει φτάσει στη βάση της υλοποίησης. Και έχουμε επίση και την ιεράρχη τη σχετική με τα απορρίμματα με τα απόβλητα, διότι κάθε κράτο μέλο υποχρεούται να εφαρμόσει αυτή την ιεράρχηση και να ετοιμάσει και επιχειρησιακά σχέδια σε σχέση με αυτό. Πάνω πάνω βέβαια, πρώτη προτεραιότητα είναι να μην έχουμε απόβλητα. Άρα, πρώτο στόχο είναι να ελαχιστοποιήσουμε την ποσότητά του. Δεύτερον, επαναχρησιμοποίηση. Τρίτον, ανακύκλωση κατόπιν ε, επαναχρησιμοποίηση με στόχο την παραγωγή ενέργειας όπως γίνεται με τους αποτεφρωτήρες και τελευταίες είναι οι χωματερές η σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη διαφέρει πάρα πολύ επομένως ξεκινούμε από τα κοινοτικά δημοτικά απόβλητα και πέρα έχουμε κάποια στοιχεία και έχουμε πέντε χώρες που έχουν σχεδόν ανυπαρξία ε, χωματερών. Δεν έχουν, δεν έχουν. Δεν έχουν πια μερικά από αυτά. Έχουν από τη φροντίδα μερικά άλλα κατέβαιναν στην ε, ανακύκλωση. Επτά κράτη-μέλη που όλα τα στέλνουν 80% συν τα στέλνουν στις χωματερές. Έχουμε βέβαια και παράμεσες ε, χωματερές και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Διότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Βλέπετε, μόνο στην κατεύθυνση πηγαίνουν τα πράγματα. Έχουν τα σχέδια, είπαμε σε επόμενε δημοσιογραφικέ πρόκειται να καλύψουμε ε, για να υποστηρίξουμε περισσότερο τις επιλογές που ακολουθούν αυτή τη λογική και φιλοσοφία. Ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση. Γιατί σήμερα ακόμα υποστηρίζουμε κάποιες ε, κινήσεις, δραστηριότητες σχετικές με την χωματερή. Ή αλλιώ θα είχαν γίνει χωματερές οι πόλεις μας. Αυτή λοιπόν είναι η αλλιως θα ειχαν γινει χωματερες οι πολεις μας. Κοιτάξτε. Δεν μιλήσαμε ακόμα για τα σκουπίδια που βρίσκονται τώρα στις χωματερές. Μάλλον η δυσκολία της ε, διαλογής είναι εμπόδιο που να ξεπεραστεί τόσο ώστε να προχωρήσουμε και κάτι να βγάλουμε και από εκεί. Πάντως ποτέ μιλάς ποτέ. Αυτό πιστεύω the story which I have explained at the beginning of how our resources have been consumed and how Οπότε θα πρέπει να δούμε το, τη διαδρομή των πόρων μας, πώς γίνεται η ανάλωσή τους, πώς ε, έχουμε φτάσει στα όρια σε ορισμένους πόρους, γιατί είτε μας αρέσει όχι. Η ανακύκλωση και αυτή η φιλοσοφία μας σε σχέση με το πόσο έχουμε τη ζωή μας. Κάποια στιγμή όλα αυτά τα πράγματα γίνουν πραγματικότητα. Άρα χρησιμοποιούμε τώρα συχνά, αρκετά, την καινοτομία. Αυτό το οποίο θα χρειαζόταν θα ήταν να στείλουμε ένα μήνυμα σαφές ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αν είμαστε ξεκάθαροι σε σχέση με αυτό, τότε είμαι σχεδόν σίγουρος ότι τότε θα πιστοτευτούν όλοι και όλα ούτως ώστε αυτό το οποίο ήταν ένταση εργασίας τώρα να πάει εκεί που θέλουμε. In the, in the resources productivity there are still major major reserves. Ε, υπάρχει τώρα για την παραγωγικότητα, βέβαια δεν υπάρχουν θέματα, υπάρχουν επιφυλάξεις και ξέρετε πάρα πολύ συχνά μιλώ σε μεγαλοεπιχειρηματίες that's exactly the right diagnosis and that... Ναι, συμφωνούν. Ναι, αυτή είναι η σωστή διάγνωση. Επομένως αυτοί που βλέπουν πιο μακριά το βλέπουν καθαρά ότι το μέλλον είναι εξοικονόμηση πηγών ενεργείας. Και έτσι οφείλεται και το περιβάλλον. Άρα λοιπόν, οι δυνατότητε που πάρουν σε με την κοινοτομία μα δίνουν το μέλλον με την τιμολογιακή πολιτική θα δώσουμε κίνητρα προς τούτο. Και έτσι θα συνδυάσουμε όλα τα μέσα πολιτική τα οποία έχουμε. Ο... Κύριε Γιόνσον, περίπου και αυτό, αυτό που είμαστε σας καλύπτει σε σχέση με το πώς θα προχωρήσουμε όσον αφορά τις τεχνολογικές μας, τους τεχνολογικούς μας πόρους, ας πούμε. Χθες Ήρθα σε επαφή με το ΣΕΦΙΚ. Ξέρετε τι είναι. Είναι αυτή η ένωση βιομηχάνων. Βέβαια σε κάθε φάση μετασχηματισμού έχουμε αυτούς που κερδίζουν για αυτούς που χάνουνε. Αλλά είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία. Γιατί έτσι Βλέπουμε τι γίνεται με αυτέ τι απέσει ουσίε, τι τοξικέ, αυτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Είναι αυτά που έχουμε συμφωνήσει τώρα. Και τώρα έχει δοθεί η ευκαιρία να έχουμε υλικά τα οποία θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Να, τι συνδυασμού θα πρέπει να κοιτάξουμε, τι συνδυασμού θα πρέπει να προωθήσουμε. Γκέρεκ, Πολύ ευστοχερό ερώτηση. Και όντως εκεί υπάρχει μια συνέπεια ότι θα θέλατε να χρησιμοποιείτε λιγότερου ενεργειακού πόρους, αλλά απ' την άλλη θέλουμε να εξωθήσουμε τις τιμές προς τα πάνω. Γιατί αυτό? Γιατί υπάρχει σπάνιση αυτών των πόρων και άρα θέλουμε με τις, με τις ακριβότερες τιμές να χτυπήσουν το καμπανάκι του κινδύνου. Εάν όμως θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα με το, με το, με το κόστο εργασία. Αυτό είναι κάτι που του βρίσκει όλου. Συμφωνούν. Είναι το μόνο που συμφωνούν όλοι, ότι είναι πάρα πολύ ακριβή εργασία στην Ευρώπη. Και επομένω θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τη φορολόγηση. Πού θα πάει η φορολόγηση, θα πάει στην εργασία ή θα πάει στου ενεργειακού πόρου. Εντάξει, έτσι γίνεται τα πράγματα πιο ακριβά, ανεβαίνει το κόστο, αλλά στέλνουμε το, το μήνυμα. Και έτσι δεν χάνουμε σε ανάπτυξη. Οπότε έτσι δεν τιμωρούμε ούτως υπήρχε την εργασία. Έτσι διατηρείται το βιωτικό επίπεδο, αυτό το οποίο έχουμε, αυτό που έχουμε συνηθίσει και που δεν θέλουμε να πέσει, να μείνει ψηλά. Όλα αυτά όπως βλέπετε λοιπόν, συντεριάζουν. Έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι το μέλλον. Έτσι είναι τα πράγματα, αλλά εμείς είμαστε οι αγγελιοφόροι, εμείς οι πολιτικοί. Το μέλλον ήδη είναι εδώ. Η ενέργεια που αναφέρατε. Η πόρη. Ε, η ενέργεια είναι. Ο βασικό ποσό, μιλούμε για αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι μιλούμε για ενεργειακή χρησιμοποίηση ενός των ενεργειακών πόρων. Να, τι εν μέρη καλύπτει αυτό το οποίο είπατε. Διότι Πάνω σε αυτό θέλουμε να επισύρουμε την προσοχή σας. Ήδη. Σήμερα έχει διαμορφωθεί συνένεση. Σε σχέση με το ότι υπάρχει σπάνιση στην ενέργεια και άρα θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη χρήση της. Ήδη έχει διαμορφωθεί στον επιχειρηματικό κόσμο συμφωνία όσον αφορά τις πρώτες ύλες ότι υπάρχει σπάνιση και εκεί ότι εάν δεν ληφθεί αυτό το γεγονό υπόψη, τότε θα του χτυπήσει πάρα πολύ σκληρά η αγορά. Όμω υπάρχουν σήμερα κάποιοι πόροι που δεν θεωρούνται ότι έχουν, ε, έχουν πρόβλημα. Αυτό όμως είναι ο για τα ψάρια. Αφού λέμε ότι έχουμε 88% υπεραλίευση. Να, τι θα πρέπει να διέπει τη διαχείριση της οικονομίας μας συνεχώς. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε και όσον αφορά τα είδατε όπως ακριβώς είπατε. Βεβαίω και το νερό είναι ένα ενεργειακό πόρο. Αλλά θυμάμαι όταν σπούδαζα οικονομικά, μου είπαν ότι είναι δωρεάν το νερό. Δωρεάν εμπόρευμα θα, θα πει εμπόρευμα που δεν έχει τιμή. Δεν, ε, δεν και τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι άλλαξαν τα πράγματα από τότε. Και το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα οικοσυστήματα, πρέπει να λάβουμε υπόψη το, το, το, το ότι η γη θα είναι πάρα πολύ σημαντικός καταλήτης στο μέλλον. Γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση και ανταγωνιστικότητα σχέση με τη γη. Οι υποδομές, η γεωργία, η ενέργεια, όλοι αυτοί ανταγωνίζονται για το ποιος θα χρησιμοποιήσει τη γη του έδαφους. Είδατε πώς φωτίζουν τα μάτια των παιδιών μα να πηγαίνουμε βόλτα στην φύση. Πόσο τα μαγεύει η φύση. Ε, καλά, ναι, όταν μεγαλώνει κανείς, χάνεται αυτή η μαγεία. Όμως, ας προστατεύσουμε τη φύση. Για το μέλλον, ο κύριο Κέλλη τώρα. Ρώτησε για τους στόχους. Νομίζω ότι οι στόχοι θα πρέπει να εξετάζονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Γιατί όσον αφορά πολύ. Για μένα είναι ένα το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Είναι γεγονό η αλλαγή του κλίματο. Εάν η απάντηση είναι καταφατική, τότε δεν υπάρχει αναλλακτική. Είναι γεγονό ότι Πώς έχουν σήμερα τα πράγματα ε, παγκοσμίω. Είναι δύσκολο κανείς να καταφέρει να πείσει όλο τον κόσμο σχετικά με αυτό. Όμω. αυτό προείπα, όμως είπαμε, αυτέ είναι οι τάσει που κυριαρχούν και θα πρέπει επί τη βάση αυτών κανείς να προετοιμαστεί γιατί συντόμω δεν θα υπάρχουν εναλλακτικέ. Ε, καλά, γιατί εμεί όμω να κάνουμε την αρχή για να μην κάνουν οι άλλοι, δεν θα σε κανεί. Μα αν δεν υπάρχει εναλλακτική. Ε, Όπω ισχύει για την αποτελεσματική χρήση τη ενέργεια, αυτό που θα είναι πιο νωρί έτοιμο. αυτός θα κυριαρχήσει στην αγορά. Αυτός θα είναι η πρωτοπορία. Βεβαίω, Μην υποτιμώ του άλλου ότι δηλαδή δεν βλέπουν αυτή την ευκαιρία για να ρίξετε μια ματιά στο πενταετές πλάνο της Κίνα, θα δείτε ότι είναι πιο πράσινο από το δικό μας και έχουν και ένα πλεονέκτημα σε σχέση με εμάς. Το είπα. Είναι διαφορά τους σε σχέση με τη δική μας κοινωνία. Εμείς έχουμε κάποια στεγανά στην κοινωνία μας. Αυτοί δεν έχουν. και οι Αμερικανοί και οι Ιάπωνες το ίδιο πρόβλημα τα στεγανά η Κίνα όμως και οι άλλες αναδυόμενες οικονομίες συνέχεια αναπτύσσονται συνέχεια επεκτείνονται οπότε και οι δυνατότητε τους προσαρμόζονται σε αυτή την τάση να και για τα πάνελ τα ηλιακά είναι πρωταγωνιστές στον κλάδο η Ευρώπη ακόμα ασχολείται με την παραγωγή, την ε, φιλοπεριβαλλοντική λογική. Άρα να δούμε πώς θα ενισχυθεί, πώς θα είναι πιο ανταγωνιστική η βιομηχανία μας. Προς τα μέσα θα πάει καλά η Γερμανία, έχουν τους στόχους όσον αφορά την κατανάλωση, το, τι παράγουν. Έχουν πάρει το δρόμο τους για τους στόχους αυτούς και εν μέρη ή εν όλο η επιτυχία της Γερμανίας έχει να κάνει με τις διαφορετικές αλλαγές που εδώ και καιρό λαμβάνουν χώρα και τους έχουν οδηγήσει στην ανταγωνιστικότητα. Να γιατί μιλάω για ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Άρα βλέπετε πως η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα. Το εξόριξη άνθρακα τώρα και τα σχετικά. Μίλησατε εσείς για το Energy Mix, το ενεργειακό μείγμα πολιτικής. Βέβαια, σε αυτό έχουν τα κράτη-μέλη διακριτική ευχαίρεια, ελευθερία επιλογής. Όμως, όχι όσον αφορά τι ανέσουμε πηγές, ενέργειας, γιατί έχουν δεσμευτεί να πάμε στο 20, 25, 15% ανάλογα με το σημείο γίνηση για κάθε χώρα. Βασικό μα προσανατολισμό αυτός, βασικό ε, τμήμα τη φιλοσοφία μας. Και τότε, θυμάμαι, ο Πίμπολτ ήταν ε, υπεύθυνο και μαζί. Θεωρήσαμε ότι αυτό είναι ένα μέσο πολιτικής που θα πρέπει να το υποστηρίξουμε, να το προωθήσουμε 6-7 πρωτοβουλίε. είχαμε το μέσο πολιτικής που αφορούσε το διοξίδιο είπαμε να, δούμε πώς θα και είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον το κάρβονο. Γιατί έγινε αυτή η μαγική στροφή από τον έδωσε ενέργειες. Δεν γίνεται έτσι όμως αυτό. Θα πρέπει να δούμε σιγά σιγά πώς θα γίνει καθαρότερο, πιο περιβαλλοντικό το κάρβονο. So, so ε, to conclude, because this is more or less everything what you θα That this cross, that this, uh, what, what actually I'm trying to work... Σκληρά προσπαθώ να δω πώς θα γίνει ολοκληρωμένη ε, πρόοδος συντονισμένη σε όλες τις πολιτικές. Εάν από την αρχή τη χάραξη μια πολιτικής δεν καλυφθεί αυτό το οποίο θέλουμε, αυτό που είναι μέρημνά μας, τότε τελικά δεν θα χρειαστεί να έχουμε κατασταλτική αυστηρή νομοθεσία. Γιατί υπάρχουν στοιχεία ότι έχει σημασία αυτό που συζητούμε για τη ζωή μας, για τις πόλεις που ζούμε. Είναι σαφέ αυτό. Η συγκεκριμένη ζωή, όταν έχει κάνει σε σπίτι του και βγάζει τα ρούχα τη δουλειά, ξέρει, ξέρει τι είναι, ποια είναι η Γι' αυτό και χρειάζεται να συνεργαστούμε. Και θεωρώ ότι υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον. Ενδιαφέρει, συμφέρει την Ευρώπη, την Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και έτσι να μπορέσουμε να φτάσουμε στους στόχους που θέλουμε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που πήραν τον λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας, για τις πληροφορίες σας. Δεν νομίζω ότι είναι η τελευταία φορά που θα συναντηθούμε για το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή μας. Γιατί η εξέλιξη όλων αυτών των στοιχείων προφανώς θα μας ε, ε, ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά όλους αυτούς τους πόρους. Οπότε θα τα ξαναλέμε και τα επόμενα, τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Ε, θα τα ξαναπούμε λοιπόν κύριε Επίτροπο, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Vážené kolegyně, kolegové, budeme tedy pokračovat v dalším... Λοιπόν, συνάδελφοι, ναι. νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 19, τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Κέντ Γιώχανσον. Κύριε Γιώχανσον, έχετε το λόγο. Uh, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, καλωσορίζω την ε, πρόταση της Επιτροπής και στην έκθεσή μου τόνισα τέσσερα σημεία. Καταρχάς η Ευρώπη θα πρέπει να αποδεσμεύσει την ανάπτυξη από την κατανάλωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να ε, βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να μειώσει την σχετική εξάρτησή της από, τους, ε, από τις εισαγωγές των πόρων. Δεύτερον, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν για να εφαρμόσουν την πολιτική. Θα πρέπει να υπάρξει πιο, πιο στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό η Επιτροπή θα πρέπει να έχει σαφείς στόχους, έτσι ώστε να μπορεί να μετράει και την επιτυχία των κρατών μελών και την πρόοδο των κρατών μελών. Επίσης, ε, ε, καλωσορίζουμε την ε, πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη μετατόπιση της φορολόγησης από την εργασία προς την κατανάλωση των πόρων και χαιρετίζουμε και την πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις επιβλαπτικές δις για το περιβάλλον επιδοτήσεις. Και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας για τη Σουηδία και το άκουσα από το Επίτροπος, εμείς ε, οι χώρες της Σκανδιναβίας έχουμε ένα δυναμικό για το πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στις ανάγκες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτες ύλες και μπορούμε να αναπτύξουμε ε, περισσότερο τον ορυκτό, τον μεταλλευτικό και τον δασικό πλούτο της Ευρώπης. Είναι η πρώτη φορά που, είμαι, που δραστηριοποιούμε στην Επιτροπή και ελπίζω να συν να συνεργαστείτε μαζί μου όπως και με την κυρία Εκ προηγουμένως. Επίσης να σας πω ότι ήταν πολύ καλή η συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές και σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα όντως είναι πάρα πολύ κρίσιμο η, η, η, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μιλάει με μία φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώχανσον. Πάντα οι σκιώδεις συγητές συνεργάζονται καλά με, τους, με τον εισηγητή. Είναι μια καλή παράδοση στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Γκέρεκ, σαν σκιώδης συγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι μια συνέχιση της, ένα είδος συνέχειας που δίδουμε στην ε, συζήτηση που είχαμε τον Επίτροπο όσον αφορά τους, ε, τις πρώτες ύλες και τους σπόρους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε <clears throat> τι μας οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση. Τρεις είναι βασικοί, βασικά οι λόγοι. Καταρχάς ότι αυξάνεται ο πληθυσμός, Ο πλανήτης μας όμως δεν διευρύνεται, δεν ε, ε, αυξάνεται, επομένως αυξανόμενος ο πληθυσμός μειώνεται το κατακεφαλήν ε, αντίστοιχο των, των πόρων. Υπάρχουν χώρες όπως η Κίνα παραδείγματος χάρη που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όσο δυνατόν περισσότερο αυτά που έχουν και να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία τους. Και η Ρωσία θα εξυγχρονίσει την οικονομία της κάποια στιγμή και θα θέλει να ε, εκμεταλλεύεται και να επεξεργάζεται τις ε, πρώτες ύλες της ε, επιτόπου, όπως κάνει και η Κίνα εξάλλου. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για να δούμε και πώς διαμορφώνεται το μέλλον και για μας. Επίσης, στο άμεσο μέλλον, αργά ή γρήγορα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να στραφούμε και σε χώρες όπως η Τουρκία, ας πούμε, η Ινδία, διότι πάρα πολλά πράγματα δεν θα μπορούμε να τα παράγουμε στην Ευρώπη. Τώρα, πώς μπορούμε να διορθώσουμε αυτά τα προβλήματα ή κάποια από αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει το θέμα της υποκατάστασης. Υπάρχει μία σειρά υποκαταστάτων για τα προϊόντα τα οποία δεν μπορούμε να παράγουμε εδώ. Η υποκατάσταση είναι ένα εργαλείο του μέλλοντος. Και προφανώς θα αλλάξουν και θα αλλάξει και η, κατανάλωση, διότι θα, θα καταναλώνουμε προϊόντα διαφορετικά που έχουν όμως την ίδια σκοπιμότητα. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εντροπία του συστήματος. Και για να λάβουμε υπόψη μας την εντροπία του συστήματος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το τρόπο με τον οποίο θα εκμεταλλευτούμε το, τις πρώτες ύλες οι οποίες εξορίσονται πώς θα χρησιμοποιήσουμε το μετάλλευμα, πώς θα χρησιμοποιήσουμε το, τελευταίο, το τελικό προϊόν κτλ. Η Γερμανία ούτως ή άλλως και αυτή την πολιτική θέλει να ακολουθήσουμε, αλλά καλό θα είναι να δούμε και ποιες ήταν οι πολιτικές των μεγάλων εταιριών τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την διασπάθηση των πρώτων υλών και εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τέλος πάντων, θα πρέπει να πείσουμε, πιστεύω, τους ε, πολίτες μας ότι η χρησιμοποίηση κάποιων πόρων θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης, Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ. Εκ μέρου του κυρίου Μαρτσινκίεβιτ θα ήθελα να μιλήσω. Ήθελα να προτείνει και αυτό κάποια πράγματα για την έκθεση. Τα οποία είναι τα εξή. Μιλάει για την ε, ανακοίνωση της Κομισιόν για την ε, καλύτερη χρήση των πόρων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ε, εισηγητή για το σχέδιο Είναι σημαντικό το Κοινοβουλίο να εμπλακεί ενεργά στην εργασία αυτή. Ε, Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε και αισιόδοξοι. γιατί αυτό που έχει σημασία είναι τελικά να αλλάξουμε το παρόν σύστημα παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα γίνει η παραγωγή και η χρήση των πόρων πιο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά και φιλική προς την δημόσια και την ανθρώπινη ζωή. Η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει κάποιους πόρους, που είναι δύσκολο βέβαια, που ήταν δύσκολο στο παρελθόν να εξαφθούν αλλά τώρα είναι, να εξορεχθούν, συγγνώμη, αλλά τώρα είναι πιο εύκολο. Οπότε είναι σημαντικό να γίνει αυτό. Δεν πρέπει να προωθηθούν τα ε, προγράμματα εξόρυξης, γιατί είναι σημαντικό. Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε όλο και περισσότερους πόρους και πρώτες σύλλες. Ε, πρέπει λοιπόν να τονίσουμε περισσότερο και την έννοια της ε, ανακύκλωσης. μιλήσατε για την Κίνα, την Κορέα. πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιους υποστηρικτικούς μηχανισμούς. Η Κομισιόν βέβαια προτείνει τους μηχανισμούς της αγοράς. Είναι σημαντικό επίσης να ε, δημιουργήσουμε μια σωστή νοοτροπία για τους καταναλωτέ. και επίσης θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην διαχείριση των αποβλήτων. Επίσης, εκμετάλλευση των ε, νέων πόρων, όπως το συστολιστικό φυσικό αέριο. Αλλά να μην ξεχνούμε και αυτούς που ήδη μας έχουν βοηθήσει, όπως ας πούμε ο άνθρακας. ας πούμε η πολύ υψηλή εκμετάλλευση του ενός πόρου που είναι κατά των περιβαλλοντικών αρχών μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να σημαίνει νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Πρέπει να δούμε και τα αισιόδοξα και τα πεσιόδοξα σενάρια που να λαμβάνουν υπόψη και την, ε, ε, ενεργειακή, και την επόδοση της ε, μεταφοράς και να εμβαθύνουμε την αναλυτική εργασία που κάνουμε. Αυτό θα πρέπει να συμβάλλει έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα για την κατανάλωση, την ε, παραγωγή και την ε, λογική χρηστή διαχείριση των πόρων. Ε, hm, ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομίλησε, οπότε να δώσουμε τώρα το λόγο στην Κομισιόν. Okay, thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον εισηγητή για το σχέδιο της έκθεσης. Ε. Ακούσαμε και τον ε, Επίτροπο, βέβαια δεν νομίζω ότι παρακολούθησα όλα όσα είπε. Πολλά στοιχεία όμως που αφορούν την αποτελεσματικότητα των πόρων εμφανίζονται και στην ε, έκθεση ε, του εισηγητή. Τα πάντα όμως πολλά μάλλον εξαρτώνται από την ε, θέληση των κρατών μελών να εφαρμόσουν ε, την πολιτική, την πολιτική που προτείνεται και στον οδικό χάρτη. Ένας από τους στόχους του οδικού χάρτη είναι να ευθυγραμμίσει τους στόχους με τα, και τα οράματα ε, που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, να, να, να ευθυγραμμίσει τους στόχους της Κομισιόν των κρατών μελών και χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως και το Κοινοβούλιο για να γίνει κάτι τέτοιο ε, καλωσορίζουμε την έμφαση που δίδεται ε, στην μετατόπιση φορολόγησης από την εργασία προς την κατανάλωση των πόρων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να έχουμε τις σχετικές τιμές ε, σε σωστό επίπεδο και επιτρέπεται και με τον τρόπο αυτό και με, την, και με τον τρόπο αυτό γίνεται και καλύτερα και η δημοσιονομική ολοκλήρωση. Επίσης ε, είναι σημαντική και σταδιακή κατάργηση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων. Σημειώσαμε τις διάφορες προτάσεις που γίνονται. Οι βασικές ε, Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τις ε, πολιτικές ανακύκλωσης ε, και υποκατάστασης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ε, θα πρέπει να περιορίσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πόρων που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη και αυτό είναι ένα στόχος ε, τον, ε, τον οδικό χάρτη και αυτό είναι ένας από του οδικού χάρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλου για τι παρατηρήσει τους. Έλα. Θα ήθελε κάποιο να προσθέσει κάτι. Ε, Πρόεδρε, Απλώς να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους και την Επιτροπή για τα σχόλια. Χαίρομαι γιατί μπορούμε να συνεχίσουμε την συνεργασία μας. Είμαστε στην Επιτροπή Περιφερειών και ήμουν και εκεί πρόεδρος της ομάδας Άλντε και πραγματικά έχω συνηθίσει ε, να συνεργάζομαι καλά με τους συνεργάτες ε, και ελπίζω ότι αυτό το κλίμα καλή συνεργασίας θα συνεχίσει και να καταλήγουμε, καταλήγουμε πάντα στην, στις καλύτερες εκθέσεις. Ευχαριστώ. Να σας πω ότι η προθεσμία για την υποβολή των ε, τροπολογιών είναι 1η Δεκεμβρίου το μεσημέρι. Ωραία. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης. Προφανώς υπάρχουν τα διάφορα, αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι. Εάν όχι, να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 29 Νοεμβρίου από τις 3 η ώρα το απόγευμα. Εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ.